Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους σας καταρχάς, σε όλους. Έχουμε πολύ σφιχτό πρόγραμμα σήμερα. Ψηφοφορίες, καλωσορίζω και ένα τηλεοπτικό συνεργείο του Κοινοβουλίου που κινηματογραφεί την κυρία ε, Λίντα Μακάβαν. Μακάβαν TV το λέτε, πώς είναι το κανάλι. Θα ήθελα λοιπόν αμέσως να περάσουμε στην πρώτη ψηφοφορία. Σας παρακαλώ. Και ζητεί το λόγο ο Κρίς Ντέιβις. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Δεν έχουμε μεταφράσεις των τροπολογιών από ό,τι κατάλαβα στις διάφορες γλώσσες. Και σύμφωνα με τον κανονισμό οι σκιώδε βέβαια εισηγητέ ε, από τις διάφορες πολιτικές ομάδες συμφωνούν με την εισηγήτρια ε, να συνεχίσουν παρόλα αυτά για λόγους που κατανοώ να, να περάσουμε σε ψηφοφορία. Αλλά μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ. Παραβιάζουμε τον κανονισμό και προχωρούμε σε ψηφοφορία χωρίς να έχουμε τη μεταφράσεις των τροπολογιών. Γιατί συμβαίνει αυτό. Wir haben, lieber Chris Davis, wir haben uns darauf geeinigt, ε, συμφωνήσαμε, κύριε Κριστέβης, όταν ορίσαμε τις ε, προθεσμίες για την έκθεση αυτή, ότι οι τροπολογίες θα κατατεθούν στα αγγλικά. Είχα ρωτήσει τότε αν διαφωνεί κανείς. Δεν διαφώνησε τότε κανείς. Και τώρα ε, μου λέει ο κύριος Κράμερ και θα του δώσω το λόγο για το ζητή ότι διαφωνεί, αλλά τότε δεν είχε διαφωνήσει κανείς. Είχαν πει όλοι θα υποβάλουμε τις απολογίες στα αγγλικά, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Κράμερ, ο οποίος κατέθεσε τις ίδιες τις δικές του τροπολογίες στα αγγλικά. Οπότε, να του δώσω το λόγο για να μας εξηγήσει γιατί διαφωνεί με αυτή τη διαδικασία τώρα ενώ η Επιτροπή είχε συμφωνήσει. Για να μην παρατηρούμε τη διαδικασία και να μπούμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Ματίας, ο κύριος ε, Κράμερ. Δεν θέλω να ε, σας κουράσω άσκοπα και να μακρηγορήσω. Θεωρώ όμως ότι ο κανονισμός είναι η βάση για την οργάνωση της κοινοβουλευτικής εργασίας. Και δεν πιστεύω ότι μπορούμε ε, όπως μας ταιριάζει, μας βολεύει, να τον εφαρμόζουμε ή όχι. Τώρα το θέμα είναι ε, ε, ζήτημα συναπόφασης, περίπλοκο, δύσκολο, χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται και κόπο για να καταλάβει κανείς τι διαβάζει και είναι από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα των βουλευτών να το πράττουν αυτό στη μητρική τους γλώσσα, αν το επιθυμούν. Μπορεί εγώ να απουσίαζα εκείνη την ώρα όταν το αποφασίσατε, το δέχομαι για αυτή τη φορά, αλλά έχω την ε, αίσθηση ότι η Επιτροπή μας δεν έχει καν το δικαίωμα να παρακάμπτει τον κανονισμό. Τι γίνεται, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετές ε, δυνατότητες ε, μετάφρασης. Να προηγείται όμως η νομοθετική διαδικασία και η συναπόφαση. Όχι επειδή ε, τίθεται σε ισχύ ο νόμος τον Ιούλιο θα πρέπει άρον-άρον να το διεκπεραιώνουμε. Δεν ανταποκρίνεται ε, αυτή η δουλειά ούτε στον κανονισμό του Κοινοβουλίου ούτε στην περιπλοκότητα του θέματος. Αγαπητέ κύριε Κράμερ, δεν καταργήσαμε τον κανονισμό. Το επιτρέπει ο κανονισμός. Θα σας πω και το πιο άρθρο. 156 εδάφιο 6 μπορεί το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να αποφασίσει ότι παρεκκλίνει. Δίνει τη δυνατότητα ο κανονισμός. Και μάλιστα την τηρούμε με ακρίβεια αυτή τη διάταξη. Έχετε τις τροπολογίες στα αγγλικά και είστε έμπειρος κι εσείς, αλλά θέλετε να ψηφίσουμε. Ε, συμφωνείτε με τη διαδικασία ή ε, θέλετε να σταματήσουμε. Λοιπόν, οι τι λένε. Να ψηφίσουμε. έχει αποφασιστεί, δεν χρειάζεται ειδική ψηφοφορία ούτε περαιτέρω συζήτηση. Να περάσουμε λοιπόν στη ψηφοφορία της έκθεσης. Είναι το σημείο 11. Τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκή Κοινότητα 726 2004 σχετικά με τη φάρμακο επαγρύπνηση. Αρχίζουμε. Η τροπολογία υπαριθμών 2 της συγκήτριας. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολόγη παριθμό 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 6 έχει αποσυρθεί 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρώτη τελική ψηφοφορία του σχεδίου έκθεσης όπως τοποποιήθηκε ηλεκτρονικά παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι. Σαρανταεπτά. Ομόφωνα. Υπέρ. Συγχαρητήρια. Δεύτερη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 50 υπέρ ουδής κατά και καμία αποχή συγχαρτήρια. Τώρα ερχόμαστε στην οδηγία. Η τροπολογία υπαριθμών 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ αυτό ηλεκτρονικά. Είναι η τροπολογική παριθμών 8, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 31 υπέρ, 13 κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Ψηφίζουμε τροπολογία υπερθυμών 9. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 Ειπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. Δηλαδή απορρίπτεται διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. Τι έγινε τελικά. Είχα μείνει στο 9 του κυρίου Κράμα. Εγκρίνεται η 4. 5 Ειπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 Ειπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. Η έξι, υπέρ κατά αποχές απορρίψετε Ερχόμαστε λοιπόν στο σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά πάντα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. 49 υπέρ. Ομόφωνα. Καμία αποχή και καμία ψήφος ε, κατά το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος τώρα και πάλι ηλεκτρονικά. Άρχιτε ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 50 υπέρ, κανείς κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια θερμά στην κυρία Μακάβαν. Μπράβο Λίντα. Und natürlich wird και φυσικά η έκθεση θα μεταφραστεί στο σύνολό της σε όλες τις γλώσσες. Έτσι ως υπόδειξη το παραλαμβάνω αυτό. Ερχόμαστε στην έκθεση του Chris Davis τώρα. Κοινή ελευτική πολιτική. Και ζητεί το λόγο ο κύριος Davis, παρακαλώ. Πολύ σύντομα. 550 ήταν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν στη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ τους και που ε, με βοήθησαν να το μειώσουμε για να είναι πιο εύχριστο. Είναι μεγάλη συνένεση μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων για τις συμβαστικές τροπολογίες. Είναι πολύ λίγες οι τροπολογίες ε, με τις οποίες δεν συμφωνώ και συνιστώ καταψήφιση γιατί δεν συμφωνώ με, με το πνεύμα τους ή του κυρίου Φερέιρα, γιατί νομίζω υπερβαίνουν το πεδίο της αλλιευτικής πολιτικής. Πριν ψηφίσουμε, ε, θεωρώ ότι θα υποστηρίξουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα τη βελτιώσουμε, θα βοηθήσουμε για να έχουμε μια εφόρο αλλιευτική πολιτική και βιώσιμη για το μέλλον. Και απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους να ακολουθήσουν ε, και να δώσουν συνέχεια ε, στις πολιτικές τους ομάδες για αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Αλίας τον Ιούλιο και στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλή δουλειά τώρα μπροστά μας όμως, είπε ο εισηγητής. Πόσες τροπολογίες κατατέθηκαν. Έχουμε 38 ε, consolidated amendments και συμβιβασμούς. Πάμε στην πρώτη λοιπόν υπέρ κατά εγκρίνεται. Η ενοποιημένη δεύτερη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημένη τρίτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα πάντα ενοποιημένη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. Η 9 ενωπημένη πάντα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. Chris Davis, ήταν μόνο ε, στα αγγλικά οι τροπολογίες. Δεν διαφωνείτε τώρα? Α, καλώς, απλώς ε, για να ξέρω. Ε, προχωρούμε. Κύριε Σδέβης επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για όλη τη δουλειά που έκανε για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη τροπολογία που πρέπει να ψηφίσουμε είναι 149 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στη συνέχεια 163 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 167 της κυρίας Γκέρλινγκ υπέρ. Κατά. Ξανά, 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επόμενη 177 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 186. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 21 υπέρ 34 κατά καμία αποχή απορρίψετε. Ψηφίζουμε τώρα λοιπόν την 190 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 191 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφέ. Θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 199. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Παρά. 39 υπέρ, 14 ε, κατά, εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13. Θέλετε έλεγχο για τη 201. Καλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ. 27 κατά. Εγκρίνεται. Τη συγκητή 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 14. Ψηφίζουμε για την 14 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 204. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 213 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 2.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 221 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 222 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές. Ξανά λοιπόν, 223 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές. Παρακαλώ ε, για το 225 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 26 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. Η 226 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 228 αποσύρθηκε. 229 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 230 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 231 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 231. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 26 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. Πάμε στην 233 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ, κατά, αποχές Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 235. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 31 ε, υπέρ, 19 κατά, 4 αποχές, κατόπιν τούτου εγκρίνεται. Δεν ήταν σαφές από εδώ, από το βήμα. 236 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηδάμε τώρα κάποιες ε, ε ψηφορίες. Ε, πάμε τώρα ε, στη 254. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 258 υπέρ κατά ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 258 υπέρ. Μάλλον σηκώστε τα χέρια. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 272 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 273 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 275 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, 281 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 292 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 300 υπέρ, κατά, Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 300 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 41. Ψηφίζουμε για την 41. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3.35 υπέρ, κατά, αποχές ε, Ψηφίζουμε, ξανά, ψηφίζουμε για την 3.35 υπέρ, κατά. Αποχές ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 3.35. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 31 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 336. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 339. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 44 αποσύρθηκε. Πάμε στην 340. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 343. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα ελέγχουμε την 343. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 24 υπέρ, 31 κατά, ως εκ τούτου απορρίπτεται. Πάμε στην 343. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Στην 345 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 348 υπέρ, κατά, αποχές, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 348. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 26 υπέρ, 28 ε, κατά, απορρίπτεται. Η 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 349 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 350 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 350 ηλεκτρονικά παρακαλώ ψήφισατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται Πάμε στη 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.63 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.71 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Η 52 εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 357 υπέρ ε, ε, κατά απορρίπτεται 388 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 390 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 391 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 393 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 394 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 395 υπέρ κατά αποχές ε, <clears throat> απορρίπτεται 398 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 399 υπέρ Εγκρίνεται 400 υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές. Μισό λεπτό ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ε, ψηφίζουμε για την 400 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 22 υπέρ, 34 κατά, κατόπιν τούτο απορρίπτεται. 401 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 402 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 403 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 404 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 404. Άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 26 ε, υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 405 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 406 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 407 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ε, θα ελέγξουμε την 407. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 26 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 420 ε, Γκέρλινγκ υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 422 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 422 ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία 25 υπέρ, 31 ε, κατά, απορρίπτεται. 4, 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 424 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 425 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, πάμε στην τροπολογία 68 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 436 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 438 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 439 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 440 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 441 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 442 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 443 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 444 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 447 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 446 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 445 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 450 παρακαλώ υπέρ 4.50. Ξανά παρακαλώ, η 450 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 451 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 453 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 455 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 456 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4,57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 458 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 459 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 460, 464, ψηφίζουμε μου, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 461 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 462 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 465 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 467 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 78 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 469 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 470 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 471 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 475 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 476 υπέρ κατά εγκρίνεται, η 477 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 478 υπέρ κατά Ξανά παρακαλώ ψηφίζουμε για την 478 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. 469 λέει ο πρόεδρος, υπέρ κατά, με συγχωρείτε, διορθώνει ο πρόεδρος, προφανώς εννοούσε την 479, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 480 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα αφήνουμε αρκετές, πάμε στην 492, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται 496 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 496 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 506 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 508 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε για την 508 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Υπέρ κατά. Αποχές. Ελέγχουμε για για την 507 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 22 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. 521 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 523 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 102 υπέρ κατά. Η 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 531 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 535 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 536 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 537 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 538 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 539 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 539. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. 22 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. Η 540 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 541 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 542 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο ε, σκεπτικό, η 106 στις αιτιολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 114 υπέρ κατά αποχές ε, το ελέγχουμε ηλεκτρονικά η 114 ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. 26 υπέρ, 28 κατά. Ε, πάμε στην 115. κατά αποχές απορρίπτεται. Η 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ μα είναι Την αφήσαμε την 120, πάμε στην 121. Ψηφίζουμε για την 121. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 123 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 124 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται η 127 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 128. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 31 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 129 ηλεκτρονικά, δεν είναι σαφές. 129 παρακαλώ, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, Έκλεισε η ψηφοφορία. 35 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Η 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και έτσι φτάσαμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία που άρχεται. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. 50 υπέρ. Καμία αποχή. 8 κατά. Θερμά συγχαρητήρια Chris Davis για την γνωμοδότησή σας. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν πραγματικά σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ και πάλι τη γραμματεία και για τις ενοποιημένες τροπολογίες. Πρέπει να σας πω ότι δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ και τους Σκιώδης και το συντάκτη της νομοδότησης και τους ε, εισηγητές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ενεργειακές υποδομές λέει εδώ. Γνωμοδότηση του κυρίου Πάβελ Ποπ. Αρχίζουμε. Είστε έτοιμοι όλοι για την ψηφοφορία. Πάμε. 28. ψηφίπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 Υπέρ της τροπολογίας 30. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε για την 30. Καλώς. Αρχή η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 18 υπέρ, 36 κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται σαφέστατα. 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 35. Έλεγχο θέλετε καλώς. Ε, Η 34. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 34. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 53 υπέρ, 5 κατά. Καμία αποχή. So, dann stimmen wir ab über 35. 35. Ψηφίζουμε τώρα την 35. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38. Υπέρ. Κατά αποχές ε, την 38 ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 35 κατά. Με μία αποχή απορρίπτεται. Η 39 ψήφι υπέρ κατά εποχές και η 39 θέλει ηλεκτρονικό έλεγχο. Δεν φαίνεται από εδώ ότι ψηφίζεται. Η 39 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 30 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Πάμε στη 41 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές έχουμε. Όχι. Απορρίπτεται. Έλεγχο γιατί 41 θέλετε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ, 36 κατά. Απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ψηφίζετε. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Ψηφίζουμε την τροπολογία 43. Ψηφί Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ούτως. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 46 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 47 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 53 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 και 58 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 57 υπέρ κατά απόχες Εγκρίνεται. Η 59 υπέρ. Κατά. άποχε, Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Dafür. 62 υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. 63 εδώ έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Ένα πρώτο τμήμα υπέρ, το βλέπετε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Enthaltung ist auch abgelehnt. Αποχές απορρίπτεται και αυτό. 64 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχο, παρακαλώ. Για την 64. Δεν το καταλαβαίνω από εδώ. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 64. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 31 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απόρριψετε. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 70 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. 71. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 77 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε 27 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται η 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 80 υπέρ. Κατά. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται όπως και 80. 82. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο όμως τμήμα, όχι το πρώτο. Α, θέλετε έλεγχο, καλώς. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι το δεύτερο τμήμα της 82. Περάσα. 30 υπέρ 29 κατά. Εγκρίθηκε. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 86 χωριστή. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές ακριβώς. Ε, θα ελέγξουμε την 90 ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 υπέρ 33 κατά απορρίψετε. 91 ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε για την 91. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 39 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Η, η 93 διορθώνει ο πρόεδρος. Η 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 100 έχει αποσυρθεί 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 επίσης έχει αποσυρθεί 103 υπέρ κατά Απόχες. Εγκρίνεται. Η 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Ε, Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 107 υπέρ Τσεκ. Για την 106. Ωραία, ας την ελέγξουμε ξανά, την 106 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 51 υπέρ, 5 κατά. Μάλιστα. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 115 γιατί δεν το βλέπω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά άποχες και αυτό θέλει έλεγχο 120 ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 24 υπέρ 34 κατά απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 καταπίπτει. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Όχι, όχι. 27 διορθώνει ο πρόεδρος. 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ 135 έλεγχο καλά. Ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist 25 ε, ε, υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά, άποχες, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Ή θέλει έλεγχο. Ας το ελέγξουμε. 142.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 Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, 26 κατά. Γκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 έχει αποσυρθεί 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά Άποχες. Δεν είναι σαφές να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ, 29 κατά, 30 μάλλον, 24 υπέρ. Κατά, απόχες. Πρέπει να τα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 24. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο για την 26. Ναι, εντάξει. Ελέγχουμε την 26. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και αν ψηφίσατε όλοι τελειώνει. 32 υπέρ, 28 κατά. Δεν κρίνεται λοιπόν. Λοιπόν, ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία τώρα για τη γνωμοδότηση αυτή. Αρχίζει τώρα, ηλεκτρονικά προφανώς. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει, πέρασε. 51 υπέρ, 3 κατά, 5 εποχές Συγχαρητήρια κύριε Παύλ Πόκ. next one. We have two amendments that were withdrawn at the last moment, so if you can use it. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, το 15, κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα των προϊόντων αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Γεια. Yeah. Όσους δεν θέλουν να συμμετάσχουν και θέλουν να συνομιλήσουν, παρακαλώ να εξέλθουν τις αιθούσεις. Και όσοι θέλουν να ψηφίζουν, ψηφίζουμε τώρα. Πρέπει να σας κάνω και μια ανακοίνωση. Οι τροπολογίες 93 και 105 αποσύρθηκαν τελευταία στιγμή. Άρα δεν θα τις ψηφίσουμε. Αρχίζουμε. 54 ψηφίπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να το ελέγξουμε για την 6. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 8 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 ε, υπέρ κατά αποχές Η 57 παρακαλώ. Κατά αποχές ε, ελέγχουμε λοιπόν την 57 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφορία. Λοιπόν, 53 υπέρ, ε, εγκρίνεται. Πάμε στην 58 υπέρ. Κατά. Ε, πολύ λίγοι σηκώσαν το χέρι. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ της 58 να σηκώσει το χέρι. Τέλεια. Κατά. Αποχές έτσι λοιπόν η 58 εγκρίνεται. 59. Με προφορική τροπολογία του συναδέλφου κυρίου Πυρίλο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, η 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 67 παρακαλώ του κυρίου Πυρίλο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 13 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 14 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 16 και η 68 ε, είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε και για τις δύο. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 19 παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 72 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Η 76 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Η 77 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Η 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 23 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Πάμε στην 78 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 24 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές, ελέγχουμε την 24 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 23 υπέρ, 32 ε, κατά, κατόπιν τούτου απορρίπτεται. Η 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η 81 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για την 81, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 81. Ψηφίσετε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 25 υπέρ, 33 κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν η 81. Η 82 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 86 καταπίπτει που ψηφίζουμε για την 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, για την 32. Ψηφίσαμε για την 32. Τώρα ψηφίζουμε για την 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 34. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, η 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 91 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Η 92 υπέρ, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος της 91 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 36 υπέρ, 21 ε, κατά, κατόπιν τούτου εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 92 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 93 την τελευταία στιγμή αποσύρθηκε. Πάμε στην 94. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι 98 και 99 ψηφίζουμε ομού, ε, υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε για την 98-99. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. 23 υπέρ, 25 κατά, κατόπιν τούτου απορρίπτεται. 100 και 102 πάλι ομού, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε και τώρα ηλεκτρονικά για την 100 και την 102. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφορία. 30 υπέρ, 26 κατά. Αυτή τη φορά εγκρίθηκε. Η 103 και για την 104 μαζί ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105 αποσύρθηκε, για την 106 ψηφίσμε. υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 109 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 109. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η 109 εγκρίθηκε ψηφίζουμε για την 107 και την... Μάλλον αποσύρθηκαν αυτές οι δύο 107 και 108. Ψηφίζουμε για τη 41. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 110. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ Ε, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 43. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για τη 43. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η 43. 24 με 33. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 112 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 51 υπέρ, 55 ε, κατά. Ε, κοιτάξτε, να σηκώνετε τα χέρια σας για να μπορώ και εγώ να βλέπω καλύτερα, λέει ο πρόεδρος. 113 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές ασαφές ψηφίζουμε για την 114 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφορία εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116-117 ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 αποσύρθηκε η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα ελέγχουμε την 46 Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 31 υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για τις 47 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, η 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε για την 4 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. Απορρίπτεται. Για την 50 υπέρ κατά, αποχές, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Για την 50 ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. 36 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Η 5 αποσύρεται, η 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι ψηφίζουμε για το σύνολο της έκθεσης. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. 53 υπέρ, κανείς κατά, τρεις αποχές. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Φεραίρα, για την έκθεση. Θερμά συγχαρητήρια. Τώρα πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ε, πρόκειται για την μεταφορά των ζώων. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, για τη γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλία, και εδώ πρέπει να σας πω ότι την τελευταία στιγμή μισό λεπτό παρακαλώ η ενοποιημένη τροπολογία υπεριθμών 1 μετατρέπεται σε συμβιβαστική τροπολογία και ψηφίζουμε ακριβώς τώρα για αυτήν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε για την 2 τη συμβαστική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε για την 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, για την 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, για την 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, για την 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, για την 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Για τη 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 9 υπέρ κατά αποχές ασαφές. Ελέγχουμε την 9 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίζουμε για την 9. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε, ψήφισαμε λοιπόν 29 υπέρ, 25 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 8. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ, κατά αποχές ε, ελέγχουμε την 11 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 29 υπέρ, 26 κατά, κατόπιν τούτου εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, ε, οριακά εγκρίθηκε. Ελέγχουμε τώρα για άλλη μια φορά ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 13. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 15 υπέρ, εγκρίνεται. Η 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 21 καταπίπτει, 29 καταπίπτει, 23 β καταπίπτει και πάμε μισό λεπτό, ε, πρέπει να ψηφίσουμε για την 23β. Ποιο είναι παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 25. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 22. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 35 υπέρ, για την 35 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 37 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, γιατί 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, γιατί 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 46 ε, υπέρ Κύριε Πρόεδρε, μόλις ε, εγκρίναμε τέσσερις νέες παραγράφους ε, που λένε Ακριβώς το ίδιο πράγμα πρόκειται για το GPS, την δορυφορική πλοήγηση και την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Και θα ήταν πολύ πιο συμπαθητικό η γραμματεία να φτιάξει μία και μόνο παράγραφο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ είμαι εισηγήτρια στην Επιτροπή Γεωργίας, θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να πράξετε αυτό που σας είπα. 48 παρακαλώ, ψηφίζουμε για την 48 υπέρ κατά, αποχές εγκρίθηκε η 46 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 50 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα λοιπόν ψηφίζουμε για την ε, γνωμοδότηση, για το σύνολο της γνωμοδότησης, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η ψηφοφορία έκλεισε. 51 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές, κατόπιν τούτου η γνωμοδότηση εγκρίνεται και σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ε, θερμά η στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ λοιπόν ε, θερμά για την ε, πολύ μεθοδική δουλειά που είχαμε. Σήμερα είναι αργία, είναι εορτάζουμε το τέλος του πολέμου. Ε, και πρέπει να πω ότι μερικές φορές ε, λόγω της καθημερινότητας ε, ξεχνάμε το τι σημαίνει αυτό στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη ζούμε 27 κράτη ειρηνικά και εκπροσωπούμε εδώ 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή σήμερα την οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να μνημονεύσουμε. Προχωράμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Και είναι το θέμα του κυρίου Πυρίλο ε, που χθε δεν το εξετάσαμε. Πρόκειται για το πρώην ε, σημείο υπαριθμών 6, ειδικέ διατάξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο... Μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος. Όχι, πρώτα η κυρία Γκροστέτ και μετά ο κύριος Πυρίλο. Πρώτα θα εξετάσουμε την έκθεση της κυρίας Γκροστέτ που έχει το πρόγραμμα για την υγεία. Είναι το σημείο υπαριθμών 17. Υγεία για την ανάπτυξη, τρίτο πολιτέ πρόγραμμα δράση στην Ευρω... Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη υγεία για την περίοδο 14 έω 20. κυρία Γκροστέτ, αγαπητοί συνάδελφε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους υπόλοιπους συναδέλφους που συζητάνε τώρα μεταξύ τους ή δυνατόν να βγουν από την αίθουσα ή να πάψουν να μιλάνε και να ακούσουν προσεκτικά την κυρία Γκροστέτ. Και τώρα θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Γκροστέτ. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους όσοι επιθυμούν να συζητήσουν, να βγουν έξω για να μπορούμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει για αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Παρακαλώ κυρία Γκροστέτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα υπενθυμίσω εντάχει τα συμφραζόμενα. στι 9 Νοεμβρίου 2011 κατέθεσε το σχέδιο κανονισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσπίζοντα έτσι το τρίτο πολιετές πλήσιο για την περίοδο 2014-2020 που φέρει τον τίτλο «Η υγεία υπέρ της ανάπτυξης». 446 ε, εκατομμύρια είναι η πρικοδότηση, του προγράμματος, 60 ε, δηλαδή περίπου κάθε χρόνο. Ο στόχος ε, του προγράμματος είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στους βασικούς τομείς όπου η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προσφέρει μια πραγματική προσθέμενη αξία στον τομέα της υγείας εγγράφεται ως ετούτο στην ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 και στοχεύει στην προώθηση της καινοτομία ως προς την υγειονομική περίθαλψη και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα αυξάνοντας την ευημερία των πολιτών της Ένωσης. Ε, συγκρίνοντας με την προηγούμενη περίοδο 2007-2013 παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση 5,7% και η συνολική πρικοδόκηση του προγράμματος θα είναι συνάρτηση των διαπραγματεύσεων που τώρα γίνονται για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, ο Πίτροπος Νταλή είχε αγωνιστεί πραγματικά για να μην γίνουν περικοπές δημοσιονομικές που θα είχαν επιπτώσει επί του προγράμματος και τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη και καινοτομία στον τομέα αυτό γιατί η υγεία δεν σημαίνει έλλειμμα. Επειδή βιώνουμε τώρα αυτή την κρίση, δηλαδή κάθε ευρώ που επενδύουμε στην υγεία ε, αποφέρει στο μέλλον και μάλιστα ε, σημαίνει εξοικονόμηση σε σχέση με μελλοντικού προπολογισμού. Ε, υπάρχει μια, ένα ισχυρό οικονομικό δυναμικό σε αυτό το πρόγραμμα. Οι εθνικέ αρμόδιε αρχέ, καθώ και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορεί, οι διεθνεί οργανισμοί, καθώ και οι κυβερνητικέ οργανώσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα τη της θα εκτελέσουν τα προγράμματα. Αυτό το πρόγραμμα Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, ούτε και αποτελεί ερευνητικό πρόγραμμα διαρθρώνεται δε γύρω από τέσσερι βασικέ προτεραιότητε. Πρώτον, ε, ε, να συμβάλλει στην δημιουργία καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγεία, Δεύτερον, να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πιο ποιοτικέ υπηρεσίε και ασφαλέστερες υπηρεσίε και καθολική πρόσβαση για όλου του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Τρίτον, πρόληψη των ασθενειών και προώθηση τη υγεία Και τέταρτον, προστασία των πολιτών σε σχέση με τι διασυνοριακέ υγειονομικέ απειλέ. Θα ήθελα να περάσω στους βασικούς προσανατολισμούς τώρα της έκθεσής μας. Αρχίσω με τον τίτλο, ε, το έχουμε ήδη ξαναπεί, «Υγεία για την ανάπτυξη». Ε, ήταν ένας τίτλος που με σόκαρε ελαφρώς ε, και προτείνω λοιπόν τροποποίηση ε, και θέλω να, ε, ο τίτλος να είναι «Υγεία και ανάπτυξη» διότι θεωρώ ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στη διάσταση, στην αναπτυξιακή διάσταση όταν συζητούμε θέματα υγείας. Health for Growth ήταν στα αγγλικά ο τίτλος ε, και κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά περιοριστικός ο τίτλος σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Λάινεν, είχε αναφέρει στον Επίτροπο Νταλή την ανησυχία μα σε σχέση με τον τίτλο και γι' αυτό το λόγο το είχαμε συζητήσει. Γνωρίζω δε ότι ο Πίτροπο Νταλή δεν είναι υπέρ τη προτάσεω μου. Παρόλα αυτά σας ε, καταθέτω αυτή την πρόταση και θα ήθελα να τοποθετηθείτε αληθεύει ε, παρόλα αυτά και μπορούμε να το ε, ομολογήσουμε, να το ε, δεχτούμε ότι είναι μοχλός ανάπτυξης η υγεία γιατί δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε περίοδο κρίσης. Εξάλλου η υγεία είναι ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ποιοι είναι οι στόχοι λοιπόν του προγράμματος. Μου φαίνεται ότι είναι προφανέ και ε, θεωρώ ότι υπάρχει και μια επιτακτική ανάγκη να αποφύγουμε πάση θυσία τη επικαλύψεις, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε με βέλτιστο τρόπο του οικονομικού πόρου που έχουμε, διότι το γνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένοι λόγω τη κρίση. και άρα θα πρέπει να προσέξουμε, να παραμείνουμε σε εγρήγορση, ούτω ώστε να μην απαριθμούμε σε ένα κατάλογο μια σειρά μέτρων για την υγεία, ε, το οποίο θα μα οδηγεί σε κατακαιρματισμό ε, στην χρήση των υφιστάμενων πόρων και άρα δεν δεν θα είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Δεν είναι ο στόχο του προγράμματο να κάνουμε ε, με ένα πλήρη κατάλογο παθογενειών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, διότι έτσι και το έχω πει σε όλου του παρισταμένου συναδέλφου, ε, ότι δεν έχει νόημα να καταθέτουμε τροπολογίε υπέρ ή κατά τη τάδε παθογένεια. Παρότι φαίνεται φυσιολογικό να το κάνουμε, δεν έχει κανένα νόημα σε σχέση με το στόχο και το περιεχόμενο της έκθεσης. Α δούμε τώρα την ε, δημοσιονομική κατανομή σε αυτούς τους τέσσερι ε, στόχους. Δηλαδή, ενίσχυση της καινοτομία, ευελτίωση της πρόσβασης ποιοτικέ υπηρεσίε υπηρεσίες υγείας, ε, ε, πρόληψη των ασθενειών και προστασία των πολιτών κατά των διασυνοριακών ε, υγειονομικών απειλών. Ε, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο καταμερισμό των κονδυλίων δεν πρέπει να παγιωθεί. Δηλαδή για κάθε έναν από του στόχου όντω θα πρέπει να έχουμε ένα κονδύλι και προτείνουμε το κονδύλι να είναι προκαθορισμένο για κάθε έναν από του στόχου. Όμω κατά τη γνώμη μου αυτό θα περιόριζε το εύρο και την εμβέλεια κάποιων προγραμμάτων. Εφόσον μιλάμε για μία σειρά ετών, Ενδέχεται να δημιουργηθούν ε, προποθέσει, περιστάσει ε, που θα μα επέτρεπαν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το περιθώριο ελιγμών και να επιδιώξουμε σε μεγαλύτερο βαθμό έναν από του στόχου, ανάλογα με τι περιστάσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ιεράρχηση ε, των τεσσάρων αυτών υποστόχων. Παραδείγματο χάρη, όταν υπάρχει μια διασυνοριακή υγειονομική απειλή, δηλαδή στόχο 4 του προγράμματο, θα ήταν πρόσφορο ίσω να έχουμε και την ανταρκή χρηματοδότηση. Θα ήταν αντιπαραγωγικό εκ των προτέρων να ε, προκαθορίσουμε αυτή την ιεράρχηση των τεσσάρων προτεραιοτήτων. Ω προ την κοινοτομία τώρα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το ρόλο που διαδραματίζει η ε, οικία βιομηχανία. Δυστυχώ, ε, ξεχνούμε ότι μέσα σε ένα φάρμακο κατά του καρκίνου έχουμε τον, το ίδιο επίπεδο τεχνολογίας όπως ένα Airbus. Δηλαδή για να περάσουμε από την ενεργό ουσία στην παραγωγή του φαρμακευτικού σκευάσματο, χρειάζεται πολύ υψηλή τεχνολογία και άρα καινοτομία παίζει καθοριστικό ρόλο. Σε σχέση τώρα με το στόχο της πρόληψης. Οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να προσδιοριστούν επακριβέστερα, ούτως ώστε να εκπονούμε αποτελεσματικότερες πολιτικές. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβανομένου και των ε, κακών διατροφικών συνηθιών που σχετίζονται με γεγονός ότι όλοι έχουμε μια σχετικά καθιστική ζωή και άρα υπάρχουν πολλές χρόνιες ασθένειες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο επιπολασμός ε, της, ε, του υπερβολικού βάρους ε, στα νέα παιδιά αναμφισβήτητα θα επηρεάσει και τις ε, καρδιαγγειακές νόσους που θα παρατηρηθούν όμως σε ε, μεγαλύτερη ηλικία στο ίδιο άτομο. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να καταπολεμήσει με πιο ενεργό τρόπο τη γύρανση του πληθυσμού και τις ε, νόσους που συνδέονται με τη γύρανση. Έτσι θα εδραιώσουμε όχι μόνο το στόχο 1, δηλαδή να έχουμε καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα υγείας, αλλά και το στόχο 2, δηλαδή καθολική πρόσβαση σε ποιοτικότερες και ασφαλέστερε υπηρεσίε και ο στόχο 3 πρόληψη ασθενειών και ε, προαγωγή πρόθεση τη ε, καλή υγεία. Έτσι θα βοηθήσουμε ε, του πολίτε από σωματική και κοινωνική άποψη να παραμείνουν ενεργοί για μεγαλύτερη περίοδο, μακρύτερη περίοδο στη ζωή του, ενισχύοντα έτσι την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ω προ του ηλικιωμένου τώρα, όχι μόνο θα του βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τι παθογένειε τη προχωρημένη ηλικία ηλικία, αλλά επίση δεν θα επιβαρύνουν ε, λόγω του κόστου κοινωνική ασφάλεια σε τόσο μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Τέλο, προστασία των πολιτών σε σχέση με τι διασυνοριακέ ε, υγειονομικέ απειλέ. Ε, ο εμβολιασμό των πληθυσμών είναι ένα βασικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο όταν ανακύπτει μια τέτοια σοβαρή απειλή. Ο εμβολιασμό μα επέτρεψε να βελτιώσουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάσταση κατάσταση υγείας σε πάρα πολλά κράτη-μέλη, όμως υπάρχουν διάφορες απειλές η ολοένα και αυξανόμενη κινητικότητα ε, των πολιτών. Επίσης, η ύπαρξη ολοένα και μεγαλύτερων ε, ομάδων που λόγω περιορισμένης πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες δεν εμβολιάζονται και επίσης ε, γίνεται δεκτή ολοένα και λιγότερο η έννοια του εμβολιασμού στον πληθυσμό. Χρειαζόμαστε ενεργότερη δράση λοιπόν ως προς τη δημόσια πολιτική εμβολιασμού, ούτως ώστε να έχουμε την βέλτιστη δυνατή εμβολιακή κάλυψη. Θέλω Θέλουμε έτσι να μειώσουμε τη θνησιμότητα που οφείλεται στι νόσους ε, μέσα από μια εντατική συνεργασία, καινοτόμε συνεργασία, κοινέ διαδικασίε ε, προγραμματισμού και σχεδιασμού και θέσπιση αποτελεσματικότερων μέτρων. Εν κατακλείδη, πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με την αξιολόγηση των υποστόχων αυτού του προγράμματο και γι' αυτό σα προτείνω να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν καταχωρηθεί στα εθνικά συστήματα υγεία μέσω των προσφορών δεύτερων δικτών, παραδείγματο χάρη ε, το ε, ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ, το προσδόκιμο ζωή των πολιτών ε, τη Ένωση και ο αριθμό των ετών υγιού ζωή. Ε, Ιδού λοιπόν θα ήθελα να σας ακούσω σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία. Γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα για τις ε, ε, τροπολογίες ε, υποφυσιολογικές συνθήκες. Έχουμε ορίσει τη 16η Μαΐου και στις 20 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Προέδρε, είμαι στη διάθεση των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφε, Και τώρα θα επιθυμούσα να δώσω το λόγο στους κοιόδης για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Έκαστος, αλλιώς δεν θα προκάνουμε. Μας έχει ξεφύγει ο χρόνος. Η κυρία Βίλμοτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Γκροστέτ για την έκθεσή της. Συμφωνούμε με πολλά από τα όσα αναφέρει. Καλωσορίζω τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι ανακουφισμένη που θα υπάρξει τουλάχιστον για το μέλλον ένα πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Ανησυχώ όμως γιατί είναι λάθος οι προτεραιότητες. Όπως είπε και η κυρία Γκροστέτ, δεν είναι το θέμα υγεία για την ανάπτυξη, είναι ανάπτυξη για την υγεία. Ε, έχουμε αναστρέψει το στόχο ο κόσμος ε, ζει την οικονομική κρίση και πολύ επώδυνα στο πετσί του, χωρίς να φταίει. Και το θέμα δεν είναι μόνο τα λεφτά. Η δημόσια υγεία υποφέρει στην Ελλάδα. 40% αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες πέρσι. Στη δική μου χώρα το ΕΣΥ διαλύεται. Περισσότερο από ποτέ τώρα χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη οι κατευθυντήριες γραμμές για το screening για το καρκίνο του μαστού και του τραχύλου της μήτρας έσωσαν ζωές γυναικών. Ε, αλλιώς ε, πολλές γυναίκες δεν θα ε, έβγαιναν με διάγνωση καρκίνου παρά ε, όταν θα ήταν πολύ αργά. Ε, επίσης ο πληθυσμός γεννάει στην Ευρώπη και θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την οδό και χαίρομαι που συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά μην κλείσουμε τις πόρτες και να αρχίσουμε νέες ε, πρωτοβουλίες τώρα. Φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει εστιαστεί υπερβολικά στον καρκίνο και στο HIV-AIDS. Στο παρελθόν έχουμε πετύχει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, δεν λέω. Αλλά ε, συμφωνώ με την κυρία Γκροστέτ και την προσέγγιση τη δεν θα πρέπει να αναφέρουμε ιδιαίτερες ασθένειες για να αφήσουμε ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Να μην έχουμε ένα μακρύ ευχολόγιο κατάλογο ασθενειών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να εστιάσουμε και να διατηρήσουμε την προσοχή μας στην πρόληψη. Πολλές είναι οι προκλήσεις για την υγεία και θα μπορούσαμε να τις είχαμε αποφύγει αν είχαμε υιοθετήσει σωστές πολιτικές. Σήμερα που είναι οικονομικά η καιρή, τα προληπτικά μέτρα θα ελαφρύνουν και το βάρος από τα εθνικά συστήματα υγείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να δούμε τη διατροφή, την άσκηση. Είναι βασική παράγοντες στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των ε, σχετιζομένων με αυτήν νοσημάτων. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα θέματα γύρω από το κάπνισμα. Έχει βαρεθεί ο κόσμος να μ' ακούει να τα λέω. Ε, περιβάλλον χωρίς καπνό, καλλιέργεια καπνού στην Ευρώπη, συσκευασία τσιγάρων κλπ. Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Ε, η καινοτομία στην υγεία, νέες ε, τεχνικές περίθαλψης, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη. Αλλά ο στόχος θα πρέπει να είναι ο υγιής πληθυσμός, να είναι υγιείς οι άνθρωποι. Δηλαδή και αυτό σημαίνει μια καλύτερη κοινωνία πιο βιώσιμη, άρα και η οικονομία πιο βιώσιμη. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με την εισηγήτρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διορθώσουμε τις προτεραιότητες. Έχουμε πολλά κοινά και νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ. Τρία λεπτά, ούτε καν τέσσερα. Τέλεια. Άλλος και Είναι η Αντωνία Παρβάνοβα, παρακαλώ, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φρανσουάζα για την έκθεσή τη, για το ανοιχτό πνεύμα και το πνεύμα συνεργασία κυρίω που τη χαρακτηρίζει. Οι φιλελεύθεροι καλωσορίζουν και υποστηρίζουν την ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντα ε, την ε, σημασία του θέματο μεσού τη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε κυρίω προτεραιότητε για τη δημόσια υγεία καθώ και του στόχου μα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστήριξε η εισηγήτρια. Όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι απαραίτητη να κάνουμε παρεμβάσεις ε, και όχι δράσεις δημόσιας υγείας ε, μόνο όταν ε, υπάρχει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να υιοθετήσει αυτή τη στάση και δεν πρέπει να μετατρέψει δηλαδή το πρόγραμμα σε ένα κατάλογο νόσων όπως μας είπε σωστά η εισηγήτρια. Η ομάδα μας ως εκ τούτου θα υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής και, τις, ε, και τη στάση της εισηγήτριας. Ε, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια ε, σημεία που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Ξέρετε, ο τίτλος σε ορισμένες γλώσσες δεν είναι καν εύληπτος ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η υγεία βιομηχανία να ε, έχει τη δυνατότητα να τονώσει την ανάπτυξη ή να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας και ζωής των ανθρώπων, δημιουργώντας έτσι ανάπτυξη, αλλά πραγματικά πρέπει να προσέξουμε για να ε, στείλουμε στο σωστό μήνυμα στους πολίτες. Σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου από πλευράς δημόσιας υγείας ε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί ως προς τον προσδιορισμό τους. Μην ξεχνάμε το θέμα στυλ ζωής και διατροφικών συνηθιών πόση σημασία έχει δηλαδή και πρέπει να συνδυαστεί η δράση μας ε, με τις δράσεις ε, άλλων ε, τομέων. Σε σχέση τώρα με την καινοτομία, ένα από τα, ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να προωθήσει την δημιουργία αποτελεσματικότερων συστημάτων υγείας, όμως δεν πρέπει να περιοριστούμε στην τεχνολογία ή σε βιομηχανικά ζητήματα. Πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία και τις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας ε, ω προ τη διαχείριση αυτών των συστημάτων και ω προ την καινοτομία που χρειάζεται κάθε σύστημα υγείας για να αναπτυχθεί. Σε σχέση τώρα με την χρηματοδότηση, την επιλεξιμότητα και την αξιολόγηση. Η ομάδα ALDE θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στα μέτρα σχετικά με την επιλεξιμότητα, καθώ και τα δίκτυα παρακολούθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σε σχέση με το mainstreaming για την ισότητα των δύο φύλων. Θα ήθελα να υποστηρίξω τι σχετικέ τροπολογίε που νέκρινε η Επιτροπή Γυναικών, γιατί ήμουν και η συγγήτρια, το λέω εν παρόδο, μπορούμε να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την ισοσκελισμένη πρόταση που αναγνωρίζει ε, την ανάγκη να βελτιώσουμε και να συμπληρώσουμε τις εθνικές πολιτικές υγείας σε ορισμένους τομείς. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Ίσως... Ε, παρακαλώ, σκιώδεις ηγητές, να εισακούονται. Αν έχετε ιδιωτικέ συνομιλίε, παρακαλώ να βγείτε τα πηγαδάκια έξω. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην άδελφο Μισελ Ριβαζή, επίσης για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Αν θέλουμε να προαγάγουμε την υγεία. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο, συμφωνώ με την κυρία Κροστέτ. Επικός απαράδεκτος όσο έχει. Δεν μπορούμε να λέμε υγεία για την ανάπτυξη, να αλλάξει, οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί. Και το τρίτο πρόγραμμα δράσης, το πολιετές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία, είναι ένας τίτλος marketing. Αλλιώς ε, ή θα έχουμε αυτό το τίτλο ή θα έχουμε ένα τίτλο πιο πιασάρικο, ας πούμε. Ε, μπορούμε να πούμε υγεία για την ευημερία, όχι υγεία για την ανάπτυξη, αν θέλετε εμπορικό τίτλο. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσουμε καλύτερα τα κριτήρια ε, κατανομής ή ανάθεσης των δικαιούχων. Δηλαδή, να μην είναι κριτές και κρινόμενοι φαρμακευτικά εργαστήρια ή δικαιούχοι, για να υπάρχει μια στοιχειώδης ανεξαρτησία. Γιατί η εγγύηση της απόλυτης ανεξαρτησίας είναι ανέφικτη. Εν πάση περιπτώσει, να το ξεκαθαρίσουμε. Για τους ειδικού στόχους τώρα. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη πτυχή για την πρόληψη. Και επίσης ε, και θα πρέπει να μπει ένα κεφάλαιο για την υγεία και το περιβάλλον. Είναι όλε αυτέ οι ασθένειε, οι χρόνιε, οι αναδυόμενε. Μιλήσαμε για την παχυσαρκία, το είπατε, επιδημίε καρκίνου, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερε στην Ευρώπη. Αν θέλουμε πραγματική πολιτική πρόληψη, κοιτάξτε τα τελευταία σκάνδαλα για τι ουσίε που προκαλούν εδοκρινικέ διαταραχέ και συνδέονται βυσφενόλοι, φθαλικέ ουσίε κτλ. με την παχυσαρκία και την εμφάνισή τη. Τι να τα κάνει μετά τα φάρμακα, στατίνε κλπ. Αυτό είναι και αμερικανική πολιτική που δίνουν σε παιδιά οκτάχρονα γιατί είναι παχύσαρκα. Εμεί θα πρέπει να φροντίζουμε να μην γίνουν παχύσαρκα τα παιδιά μα όχι να κυνηγάμε, του δίνουμε φάρμακα. Υγεία και περιβάλλον λοιπόν. Κάτι άλλο που μου λείπει και είναι σημαντικό. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις εναλλακτικές και συμπροματικές μεθόδους προς την κλασική υγεία. Όλο μας λένε για φάρμακα, για περίθαλψη νοσοκομιακή κτλ. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το πρόγραμμα για να τις προαγάγουμε ταυτόχρονα για ένα σύστημα υφόρο θεωρώ ότι εάν η καινοτομία βασίζεται μόνο στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είναι πρόβλημα, γιατί είναι πολύ συχνά πανάκριβα και δεν απαντά αυτό αυτόματα ή αναγκαστικά στις ανάγκες μας. Και θα πρέπει να αξιολογήσουμε και εκεί τις εναλλακτικές προσεγγίσεις. Για τους δείκτες. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε ε, δείκτες ακριβώς για την αξιολόγηση, αλλά θα πρέπει τα κριτήρια για την αξιολόγηση να είναι όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά για να δούμε αν φτάσαμε στους στόχους μας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στο ε, ε, όρο ευημερία, τι σημαίνει ευημερία που σας είπα, θέλουμε να βάλουμε στον τίτλο. Αν παραμείνουμε στο ποσοστό, πόσα εμβόλια πουλάμε, πόσα φάρμακα πουλάμε, τι νοσοκομεία έχουμε, με τι εξοπλισμό, αλλά η ευημερία μπορεί να είναι και η ευζοία πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται την υγεία του, ε, σύμφωνα με την, τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και για το τέταρτο στόχο, εγώ δεν πιστεύω στο μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού, ακόμα και διασυνοριακά. Το είδαμε στη γρήπη τα 1 1 ε, υπάρχουν ε, παρενέργειες και δεν θα πρέπει πάντα να θεωρούμε ότι βρήκαμε μια πανάκια που θεραπεύει τον κόσμο. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρος. Ο Ρέστε Ρώση, παρακαλώ, σκιώδης και αυτός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή μας παρουσίαση. Είναι μια πολύ σημαντική διάταξη, διότι ε, εξετάζει τις ε, δυνατότητες οικονομικές των κρατών μελών. Ε, τα λίγα αυτά κονδύλια που υπάρχουν ε, δεν είναι πάρα πολλά. Είναι κάτι πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που πρέπει να διαιρεθούν σε 28 κράτη. Δεν μιλάμε για μεγάλα ποσά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι και αυτό. Είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική συνεισφορά. Και μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Ένα τομέα που ενδιαφέρει όλου μα. Γιατί καταρχήν, α μην ξεχνάμε ότι όλα τα κράτη έχουν προβλήματα στον τομέα τη ε, περίθαλψη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό η συγγήτρια να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στο δικαίωμα των ασθενών να έχουν ίση μεταχείριση, ίση θεραπεία. Και βεβαίως πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη η ίδια σημασία τόσο στους ε, ηλικιωμένους όσο και σε αυτούς ε, που είναι σε μονεκτική θέση γιατί ε, επειδή ζουν απομακρυσμένοι δεν έχουν την διαμεταχείριση ίσως θα μπορούσαν μέσω της ηλεκτρονικής πρόβληψης ή θα μπορούσαν οι γιατροί να μεταβαίνουν επί τόπου αλλά ας μην ξεχνάμε τον κόσμο της αναπηρίας που αφορά και τους νέους. Οι ανάπηροι πολλές φορές έχουν πρόβλημα να μετακινηθούν και να μεταβαίνουν στα δικαστήρια κατόπιν. Ε, και οι σπάνιες ασθένειες ε, και εκεί οι ασθενείς ε, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τα φάρμακά τους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι θα καταθέσω τις σχετικές τροπολογίες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι δικαιώματα έχει ο πολίτης, αλλά ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και ε, να ε, γνωρίζουμε και τις ηθικές υποχρεώσει και υποχρεώσει από πλευράς του πολίτη. Ε, η δωρεά οργάνων, η αιμοδοσία. Θα πρέπει και ο πολίτης να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του αλλά και για όλα αυτά που θα μπορούσε να κάνει για να βοηθήσει τους υπόλοιπους. Και όχι και με μεγάλη προσπάθεια γιατί παραδείγματος χάρη η αιμοδοσία δεν είναι και κάτι το φοβερό. Ας έρθουμε τώρα στα θύματα. Και εδώ σκοπεύω να καταθέσω μια τροπολογία με την έννοια ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι παραπάνω στα άτομα που την χάνουν ε, θεραπείες. Γιατί πολλές φορές ε, άτομα που μπαίνουν σε θεραπεία εξελίγονται, εξελίσσονται σε θύματα. Πάνε για να πάρουν αίμα και ε, προσβάλλονται από ιούς, ακόμα και θανατηφόρους. Ή εμβόλια που και αυτά δημιούργησαν τεράστια προβλήματα γιατί ήταν άτομα που από μικρά παιδιά ήταν αλλεργικά αλλά δεν το γνώριζαν. Βελτιώνει την κατάσταση αλλά ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά και πρέπει όλα αυτά να τα προσέξουμε. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι μια έκθεση που μπορούμε να την ε, στηρίξουμε. Ε, επαναλαμβάνω, ε, η, τα κονδύλια για τα οποία μιλάμε δεν είναι τεράστια, αλλά κάτι είναι και αυτά. Πρόεδρος, έτσι λοιπόν κλείσαμε τον κύκλο των σκιωδών εισηγητών και τώρα θα ήθελα να δώσω στους επόμενους ομιλητές που θα ακολουθήσουν. Ε, αν διάβασα τα ονόματά τους, δεν ξέρω αν τα ακούσατε και αν παρέλειψα κάποιον ομιλητής. Εσείς συμπεριλαμβάνεστε στον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Χρυσόγελος σας ανέφερε. Και θα ήθελα τώρα να περιορίσουμε το χρόνο σε 2.30, 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Πρώτος ο κύριος Λίζα και μετά ο κύριος Πυρέλο ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά την Φρανσουάζα Γκροστέτ για τη δουλειά της Νομίζω ότι η δουλειά της ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και επίσης ε, και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει τώρα να κάνουμε διαγωνισμό για το ποια ασθένεια οφείλουμε να φέρουμε και ποια όχι. Να το δούμε λιγάκι το όλο θέμα κάτω από ευρύτερο πρίσμα. Πρέπει να σας πω, χαιρετίζω ανεπιφύλακτα το να αλλάξουμε την επικεφαλίδα. Γιατί όταν κάποιος έχει γενέθλια ή την πρωτοχρονιά, ε, τότε κυρίως έχετε κανείς ε, υγεία υγεία. Ε, ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η εποχή που ζούμε. Ε, δεν αισθάνεσαι όπως κανένα που να εύχεται την πρωτοχρονιά. Εύχομαι ανάπτυξη σου, εύχομαι να είσαι και εσύ μέσα σε αυτό τον κύκλο της ανάπτυξης. Ε, ξέρω λοιπόν γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε την ε, πρότασή της ε, ως τη διατύπωσε ο Επίτροπος, μας το εξήγησε. Εμείς όμως δεν είμαστε η Επιτροπή, εμείς είμαστε οι αιρετοί εκπρόσωποι του λαού και θα πρέπει να του παρουσιάζουμε, παρουσιάζουμε τους πολίτες αυτά που, του, που τους είναι σημαντικά. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηρίξουμε όλη αυτή τη βιομηχανία της υγείας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες δυνατότητε να προάγουμε την υγεία στην Ευρώπη. Δεν πρέπει απαραίτητα η υγεία να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός τομέα. Ε, πολλοί θα διορτηθούν ε, γιατί δεν παραμένουμε στα παλιά στο Health Action Program. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον αυτό να το συζητήσουμε και μετά να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι θεσμοί ίσως η πρόταση της ε, Φρανσουάζ να αποτελεί συμβαστική πρόταση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε, θέματα που έχουν ε, ευρωπαϊκή υπεραξία, σε θέματα που δεν μπορούν να τα επιλύσουν μόνα τους ε, τα κράτη-μέλη. Οι ασθένειε, πράγματι, εκεί χρειαζόμαστε κοινή δράση ή το θέμα των παιδικών νόσων, κυρίως όταν τα παιδιά ε, νοσούν βαρέως. Εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι ε, ασχολούνται με το θέμα των πρόωρων τοκετών. Και νομίζω ότι ε, θα πρέπει ή μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ αν γίνουν γνωστά αυτά τα οποία παραδείγματο χάρη πράττει η Πορτογαλία στον τομέα αυτό. Ο κύριος Πυρέλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή λοιπόν υπάρχουν περιορισμένοι πόροι και αυξάνονται όλο και περισσότερο οι ανάγκες στον τομέα της υγείας, αυτό το πρόγραμμα υπέρ της ανάπτυξης, ακόμα και εάν είναι ε, φιδωλά πρικοδοτημένο, μπορεί παρόλα αυτά να προσφέρει ε, προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που κατατέθηκε για μένα είναι αποδεκτό. Πρέπει βέβαια την προσοχή μας να την εστιάσουμε σε ένα θέμα το οποίο δεν διευκρινίζεται απόλυτα σε αυτή την πρόταση κανονισμού. Αναφέρομαι στην πρόληψη που συνδυάζεται με την φυσική υγεία ε, των πολιτών μέσα από προληπτικά μέτρα που συνδυάζονται με δράσεις που έχουν σχέση με την καλή φυσική κατάσταση μπορούμε να περιορίσουμε την ε, ε, μετάβαση την διακομιδή στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια βάση για ένα δυναμικό μοντέλο που θα αφορά ε, τον τομέα της υγείας και εκεί θα μπορούμε να έχουμε παρεμβάσεις για όλη τη διάρκεια της ε, ζωής ε, των ανθρώπων. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο θα βασίζεται στην εξειδίκευση της ε, τεχνολογίας και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και στην πρόληψη. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου του 2010. Ε, αναφέρομαι και πάλι στις εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως επίσης και στην δυνατότητα πρόσβασης στις υγείες αυτές κυρίως όσον αφορά τον τριτογενή τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος για δυόμιση λεπτά ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα γενικά να πω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Συγχαρητήρια στην κυρία Κροστέτ ε, για την καταπληκτική της εργασία. Πιστεύω ότι γενικά οι υγειονομικές τάσεις και η εξέλιξη της υγείας δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών, τα φάρμακα είναι όλο και πιο ακριβά οι δομές ε, των δαπανών και του κόστους αμφισβητούνται γιατί τα κράτη-μέλη ανασυγκροτούν τα συστήματα υγείας λόγω έλλειψης ε, οικονομικών πόρων κτλ. Στην τελευταία διάσκεψη που διοργάνωσε η Επιτροπή, η υγεία ορίστηκε ως προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και για την ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ πρόσφορο. Χρειάζεται αλήθεια ε, προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό είμαι απολύτως υπέρ της έμφασης που δίνει η παρούσα έκθεση στην πρόληψη. Εκεί αφιερώνεται ένα 3% των κρατών μελών στην πρόληψη. Μόλις 3% του ΕΕΠ αφαιρών, ή του, του προπολογισμού. Είναι πολύ μεγάλο σφάλμα και θα πρέπει να αυξηθεί οπωσδήποτε. Ελπίζω να βοηθήσει και το πρόγραμμα αυτό προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης χαίρομαι που αναφέρεστε στην ε, να συγκρότηση και μεταρρύθμιση των ε, συστημάτων υγείας. Αυτό μόνο σε κεντρικό επίπεδο μπορεί να συντονιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ανισότητες στις χώρες μέλη αναλυθούν θα πρέπει να αποφασιστεί αυτό πανευρωπαϊκά. Εκείνοι που πλήττονται όμως από αυτές τις ανισότητες είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες και ασθενείς. Ακούσαμε επίσης για τη γύρανση. Ε, είναι ένα φαινόμενο που θα οξύνεται συνεχώς. Και θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας όχι στη θεραπεία όπως είπα και προηγουμένως αλλά στην πρόληψη. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και από εκεί να αναζητήσουμε την καινοτομία. Άλλο θέμα. Ενίσχυση των συστημάτων διαπαιδαγώγησης των ασθενών για τα ιατρικά αυτά ζητήματα ή του πληθυσμού. Έχει γίνει δουλειά ήδη, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή για να καταλήξουμε σε ένα σύστημα ιατρικών δικτών σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο σε ορισμένα. Γιατί αν δεν έχουμε ένα σύστημα δικτών δεν θα μπορέσουμε να μετρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα. Και ένα τελευταίο και τελειώνω. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους δείκτες που αξιολογούν ε, την ε, αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και τη, κατά πόσο ε, ενεργών. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, για δύο μισή λεπτά και πάλι, η κυρία Ροτ Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μερικές μικρές παρατηρήσεις στην και πάλι φυσικά πολύ καλή έκθεση της κυρίας Κροστέτ που είναι η δήμον σε θέματα πολιτικής υγείας και ό,τι πιάνει πραγματικά το βγάζει τέλειο. Έχω πολύ μικρά σχόλια για το περιεχόμενο και κάποιες επιφυλάξεις. Τα σχόλια. Για παράδειγμα, στην τροπολογία παριθμών 20, η κυρία Γκροστέτ ε, αναφέρεται σε χρόνια νοσήματα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ενιαίο ορισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ισχύει παντού ο ίδιος για τις χρόνιες νόσους. Καλό και σωστό είναι να αναφέρονται με μονομένα ίδια ασθενειών όπως είναι η καρκίνη, αλλά από την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου λείπει η αναφορά σε νευρολογικές παθήσεις ή παθήσεις του εγκεφάλου. Στην τροπολογία της υπαριθμών 15 τα λέει αυτά η κυρία Κροστέτ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το ενισχύσουμε. Γιατί το πρόβλημα και τα προβλήματα στο μέλλον που θα έχουμε μπροστά μας είναι κυρίως οι νευροεκφυλιστικές νόσοι και γενικά νοσήματα του εγκεφάλου και νευρολογικά. Αυτό όμω είναι για μένα λεπτομέρειε. διότι φοβούμε ότι όλοι εμεί εδώ σκοτωνόμαστε στη δουλειά για κάτι το οποίο τελικά δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Θέλω να θυμίσω σε όλους μας τι έγινε με την νομοθεσία για τη διασυνοριακή ε, φροντίδα υγείας και περίθαψη. Τα κράτη-μέλη εκεί δεν ήταν καν πρόθυμα ότι για μικρά θέματα, όπως είναι κοινά κέντρα ενημέρωση, ας πούμε, να συμφωνήσουν ε, για να έχουμε ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ε, με νόημα είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος Πέτερλε. Να αυξηθεί το ποσοστό που αφιερώνουν τα κράτη-μέλη από το ΑΕΠ στην ε, πρόληψη γενικά στην υγεία. Θα πρέπει να αυξηθεί αυτό που είναι ε, πρόθυμα τα κράτη-μέλη να επενδύσουν για τους πολίτες τους τους ίδιους άνδρες και γυναίκες. Είναι κλάσμα των όσων δίνουν για τις υποδομές των μεταφορών. Κλάσμα, ακόμα και αν φαίνεται διαφορετικά σε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία. Και είναι ντροπή αυτά που προσφέρουν στους πολίτες και, και πρόκληση και ύβρις και ε, είναι απορίας άξιο γιατί δεν έχει ξεσπάσει επανάσταση στους δρόμους και από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Και αν δεν καταφέρουμε στην πρόταση αυτή να υποχρεώσουμε σαφέστατα τα κράτη-μέλη, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο, ας το συνδέσουμε και με ε, τις πληρωμές από τα διορθωτικά ταμεία ή με σαφείς στόχους. Αλλιώς ε, αυτά τα λέμε εμεί ωραία και καλά, αλλά δεν γίνεται πραγματικότητα. Ευχαριστώ για τα μισή λεπτά. Το λόγο τώρα έχει ο κύριο Χρυσόγελος Μικρόφωνο κύριε Χρυσόγελο. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να βάλω και μια άλλη διάσταση που είναι εξόχως σημαντική σήμερα στην εποχή της ε, αυστηρής λιτότητας αυτό που βλέπουμε είναι ότι ε, επικεντρώνεται πάρα πολύ η πολιτική στην Ελλάδα ιδιαίτερα και στις άλλες χώρες, αλλά από την Ελλάδα που ξέρω πολύ καλά, σε περικοπές των συστημάτων υγείας και δεν δίνεται καμία έμφαση σε δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υγεία, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν και στην ε, βελτίωση των οικονομικών ε, της υγείας. Όπως είπε προηγουμένως και η συγγήτρια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό, θα μπορούσαμε να πετύχουμε βελτίωση των οικονομικών με έμφαση σε προγράμματα πρόληψης. Αυτό, να σας φέρω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου. Επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι καρκίνοι του πνεύμονα, αυτό έχει εκτοξεύσει τις δαπάνες ε, στη νοσοκομιακή περίθαλψη. Επίσης προβλήματα υπάρχουν ε, λόγω της αλλαγής του τρόπου ζωής. γενικά μέχρι τώρα ε, προσοχή είναι στο τέλος της αλυσίδας εκεί που η περίθαλψη είναι πολύ ακριβή η νοσοκομιακή περίθαλψη στα φάρμακα ενώ θα έπρεπε να επενδυθούν χρήματα στην αρχή στην πρόληψη. αυτό θα βελτίωνε και την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και τα οικονομικά των δημόσιων συστημάτων. επομένως νομίζω ότι αν κάτι μπορούμε να περιμένουμε από μια τέτοια στρατηγική για την υγεία είναι να είναι στρατηγική για την υγεία για την βιώσιμη ευημερία όχι ε, να στοχεύει μόνο στα οικονομικά ή μόνο στα θέματα της ανάπτυξης. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης στην εποχή της λιτότητας ε, ένας από τους τέσσερις βασικούς ε, άξονες του, της έκθεσης που το τονίζει είναι η πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία εξαιτία τη ανεργία, εξαιτία των περιοριστικών πολιτικών μένουν εκτό συστήματο υγεία. Δηλαδή και δεν έχουν εισοδήματα αλλά και μένουν εκτό του συστήματο υγεία και δεν έχουν την πρόσβαση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης να βάλει ορισμένες αυστηρότερες προϋποθέσεις ακόμα για περιοχές όπως είναι οι νησιωτικές οι ορεινές περιοχές που δεν έχουν καν στοιχειώδη ε, πρόσβαση σε αισθήματα υγείας. δεν μιλάμε μόνο ε, για ανθρώπους που ε, είναι πολύ στο περιθώριο της κοινωνίας αλλά και κανονικές κοινωνίες όπως οι νησιωτικές σήμερα έχουν πολύ μεγάλη έλλειψη. Σας αναφέρω πολλά νησιά τα οποία είναι και τουριστικά στην Ελλάδα που δεν έχουν καν γιατρό και οι άνθρωποι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για να έχουν ιδιωτική περίθαλψη ταξιδεύοντας πολλές ώρες και δαπανώντας πολλές μέρες από την εργασία τους ή από την καθημερινή τους ζωή. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε στην έκθεση και τέτοια θέματα. Και κλείνω με ένα σημαντικό. Η, απο την καθημερινη του ζωη αρα θα πρεπει να προσεξουμε στην εκθεση και τετοια θεματα και κλεινω με ενα σημαντικο η προστασία ε, σε σχέση με υγειονομικέ απειλέ ε, από διασυνοριακέ μετακινήσει. Εδώ επειδή πολλέ φορέ λαϊκίστικες δυνάμει, και όπω είδατε και στη χώρα μου ακροδεξιέ δυνάμει, πατάνε πολύ στο θέμα αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πολιτικέ συνεκτικέ και σε αυτό το θέμα. Δηλαδή η σωστή οργάνωση τη πρόληψη, η πρόσβαση μεταναστών σε συστήματα υγεία αξιοποιώντας ευρωπαϊκού πόρου, θα μπορέσει να στερήσει επιχειρήματα από ακροδεξιέ και λαϊκιστικέ δυνάμει γιατί θα βελτίωνε ε, τα συστήματα υγείας και για τους ε, ντόπιου και για τους μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Και τώρα η Φρεντερή Κρίς για μισή λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τα είπαμε όλα ή σχεδόν όλα, οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Φρανσουάς ε, Γκροστέτη. Ε, το είπε η Ντάγμαρ ότι είναι πολύτιμη η εμπειρία που έχουμε σε αυτό το φάκελο. Εγώ θυμάμαι πόσες ώρες περάσαμε με τον καθηγητή Τρακατέλη να συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων, ε, ειδικότερα για τον τίτλο, ε, ε, ήδη τοποθετήθηκαν οι συνάδελφοι, είναι με σημασιολογικό ή ορολογικό το θέμα. Αυτό που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει ω μήνυμα προς τους πολίτες είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί για τα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι μάλλον έτσι λίγο παγωμένοι, α του πω έτσι όλοι και θα Μιλάμε χρηστικά όταν χρησιμοποιούμε τέτοιο τίτλο. Υπάρχει, υπάρχουν υπονοούμενα. Νομίζω θα παρεξηγηθούμε άμα διατηρήσουμε αυτό το τίτλο. Ο Επίτροπος Νταλή ήδη αποφάνθηκε. Θα πρέπει να, ε, σε κάθε περίπτωση να τροποποιήσουμε τον τίτλο. Ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια ως προς την ε, καινοτομία. Ε, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό τον ε, περιραίοντα φόβο και το δισταγμό. Ε, υπάρχουν πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας, της γενετικής και θα πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτήν την νέα πορεία μέσω από το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα αλλά και μέσω αυτού του προγράμματος για την υγεία να ενισχύσουμε την έρευνα. Συμφωνώ με τον κύριο Ριβαζή, δηλαδή την κυρία Ριβαζή, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν για την έρευνα Εξίσου σημαντικό πολιτικό μήνυμα είναι να δείξουμε ότι υποστηρίζουμε τα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας. 10% περίπου του ΑΕΠ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού και ακούσαμε πολλά για τις ε, εναλλακτικές ε, θεραπείες, αλλά πάντως η υποστήριξή μας για τους βασικούς ε, τομείς της υγείας πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ας αφήσουμε τώρα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα ευχολόγια με τις ασθένειες. Πρέπει να δράσουμε εκεί που προσφέρουμε μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία Ω Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουμε τα προηγούμενα δικά μα προγράμματα κατά πολέμηση της κατανάλωση καπνού, αλκοολούχων, ποτών για την παχυσαρκία. Αυτά από πλευρά πρόληψη είναι απαραίτητα, υποστηρίζονται και τους στόχους της ε, κυρίας Γκροστέτε για το γύρανση, κάτι που απειλεί κάθε έναν και σε συνδυασμό με αυτό φυσικά και τις νευροεκφυλιστικές ενώσους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να σε ενοχλήσω βέβαια γιατί φαίνεστε απασχολημένος. Uh, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Γκροστέτ. Είναι πληρέστατη η πρόταση που μας καταθέτει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής ε, που ε, εξέφρασαν την άποψή τους. Από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνουμε μεγάλη ικανοποίηση ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη συνένεση ως προς την ανάγκη να θεσπιστεί το πρόγραμμα και ως προς τους πρωταρχικούς του στόχους η υγεία των πολιτών ε, ως προς τις βασικές προκλήσεις ε, που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε στην Ένωση. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια βασικά ζητήματα που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Όταν μιλάμε για την υγεία, για την ανάπτυξη και το σχετικό πρόγραμμα, βασιζόμαστε στην εμπειρία μας. Είναι η τρίτη εκδοχή, η τρίτη διασκευή του προγράμματος. Έχουμε μια ε, εμπειρία δεκαετή με τέτοια προγράμματα υγείας. Λοιπόν, αυτό το νέο πρόγραμμα θα βασιστεί, θα εδραστεί στην εμπειρία εμπειρία των ε, παρελθόντων προγραμμάτων ε, και θα ανοίξει νέους ορίζοντες αλλά και νέες προκλήσεις. Προσπάθησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί σε αυτό με στην ε, πρότασή της. Είναι εξίσου σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τι μπορούμε να επιτύχουμε με, να, τι είναι ρεαλιστικό ως προς τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων ε, στον ε, τομέα της πολιτικής υγείας και ως προς ε, το μέγεθος του προϋπολογισμού. Είναι ένα πρόγραμμα μόχλευσης, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όπως και τα προηγούμενα, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, γιατί είναι και πολλοί άριθμοι, μην το ξεχνάμε στον τομέα αυτό, να τους υποστηρίξει τη δουλειά που κάνουν. Η επιτυχία ή η αποτυχία λοιπόν του προγράμματος θα πρέπει να αποτιμηθεί σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο διευκολύνει τις δράσεις των εμπλεκομένων φορέων και την επίσπευση ή όχι της δικής τους δράσης. Ως προς τις επιμέρους δράσεις προσπαθήσαμε να τονίσουμε ότι ακριβώς αυτό επιδιώκουμε και εμείς. Ε, Δεδομένα των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων, ε, τελικά πόσο χρήσιμο θεωρούν ότι είναι αυτό το νέο μας πρόγραμμα για να μπορέσουν να επιτύχουν τους πρωταρχικούς τους στόχους. Είναι ένα μεσαίου μεγέθους πρόγραμμα ε, ως προς τον προϋπολογισμό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αναγνώρισαν και οι συνάδελφοι και έχουμε πολύτιμη, ξαναλέω, δεκαετή εμπειρία ε, από την οποία μπορούμε να μάθουμε πολλά. Θα ήθελα τώρα ε, να σχολιάσω το θέμα του τίτλου. Σχεδόν όλοι οι προλαλήσαντες ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα. Ε, ίσως είναι θέμα κατανόησης. Ε, θα ήθελα να σε εκθέσω την άποψη της Επιτροπής. Δεν είναι ακριβώς αυτός καθ' αυτός ο τίτλος που έχει την ε, μεγαλύτερη σημασία, αλλά μάλλον ή, το πνεύμα με το οποίο επιλέξαμε αυτό τον τίτλο. Ο στόχος δεν είναι να θεσπίσουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα και σε καμία περίπτωση η υγεία δεν είναι υποδεέστερη και δεν ε, γράφεται σε μια γενικότερη οικονομική ατζέντα. Δεν ήταν ουδόλως η πρόθεσή μας. Αντιθέτως, ε, θέλαμε να περάσουμε το εξή μήνυμα. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για την υγεία. Όπως λέγαμε και στην Ευρώπη 2020 και το σχετικό έγγραφο προωθούμε ένα νέο όραμα για την Ευρώπη. Θέλουμε να επικρατήσει δικαιοσύνη για όλους και να είναι αλληλέγγυα η οικονομία. Οπότε όλα αυτά τα υπονοούμε μέσα από τον τίτλο. Επίσης ε, θέλουμε στην καρδιά του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης να βρίσκεται η υγεία και πιστεύουμε ότι αυτό ε, είναι και η επιθυμία των πολιτών. Όταν μιλάμε λοιπόν για την υγεία, για την ανάπτυξη, δεν ε, κρίνουμε φυσικά τη χρησιμότητα της υγείας επειδή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και διπιωτικές, αλλά το παραγωγικό εργατικό δυναμικό, ο παραγωγικό πληθυσμό που δύναται να μετάσχει σε οικονομικές δραστηριότητες και ε, χρειάζεται ε, εξασφαλισμένη, κατοχυρωμένη πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίε υγεία. Ε, έτσι αντιλαμβανόμαστε εμεί την ανάπτυξη σε συνάρτηση με την υγεία στην επόμενη περίοδο. Λοιπόν, έχουμε την πρόθεση να απομακρυνθούμε από την προηγούμενη έννοια τη υγεία ότι είναι ένα άχθο, συνεπάγεται μεγάλο κόστο. Δεν είναι μόνο αυτό η υγεία, είναι βασικό ε, θεμέλιος λίθος, ε, αν θέλετε, για, του, της κοινωνίας και του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης. Ε, αντιλαμβάνω πόσο δύσκολο είναι να περάσουμε όλα αυτά τα σύνθετα νοήματα μέσα από τρεις λέξεις ε, του τίτλου συγκεκριμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή ήταν η πρόθεσή μας ε, και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από όλε τι επενδύσει που μπορούμε να κάνουμε η υγεία είναι η σημαντικότερη επένδυση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίοδο κρίση. Σε σχέση με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τώρα να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα διότι απασχολεί του συναδέλφου από ό,τι άκουσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τέσσερι βασικού και συγκεκριμένους στόχους. Όλοι είναι εξίσου σημαντικοί. Αν δεν ήταν σημαντικοί, δεν θα τους απαριθμούσαμε στον κατάλληλο και ούτε και θα του αναφέραμε στην πρότασή μα. Όμω ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι στόχοι ε, σε προηγούμενα χρόνια έχουν ήδη επιδιωχθεί. Δηλαδή, τρόπον την να βασιζόμαστε στην παρελθούσα εμπειρία και γνώση ε, σε ορισμένου τομείς, ε, όπως οι υγειονομικές απειλέ, είμαστε σε φάση παγιοποίηση της παγιοποίηση ε, των προηγουμένων ε, θετικών αποτελεσμάτων. Σε άλλους τομείς ε, βέβαια τώρα ξεκινάμε και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς για πολύ ειδικά ζητήματα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά είδη επενδύσεων που είναι απαραίτητα στον τομέα αυτό. Υπάρχει επίσης μεγάλη ευελιξία, διότι υπάρχει η προγραμματική περίοδος χρηματοδότησης αλλά και άρα χρειάζεται πολυετής προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης ενδέχεται να ανακύψουν προτεραιότητες αναχρονική στιγμή, αναχρονική περίοδο. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο ε, ε, ο εκπρόσωπος της Δανικής Προεδρίας έχει ζητήσει το λόγο ή εκπρόσωπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω. Μπόρεσα να συμμετάσχω στη σημερινή ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη. Εξ ονόματος της ε, Δανικής Προεδρίας ε, και της Προεδρίας της οικίας ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Θα έλεγα σε ένα πρώτο στάδιο ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, είναι σε πλήρη εξέλιξη και άρα δεν θα μπορέσω να μπω σε λεπτομέρειες όμως. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ε, αναφερθώ σε κάποια στοιχεία της ε, πρότασης. Ε, η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας και στις 22 Ιουνίου αναμένεται να εγκρίνουμε τη θέση μας ως προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από πλευρά Συμβουλίου Προσβλέπουμε με ανυπομονησία στην επικοδομητική μελλοντική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα εργασία ισορροπημένο που να προσφέρει προσθεμένη αξία και για του πολίτε και για τα συστήματα υγεία. Ε, σας ευχαριστούμε και εν τέλει ακούσουμε και την συγκίτρια για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν ε, και ε, είμαι πεπισμένη, λοιπόν, έχοντας ακούσει τις παρεμβάσεις, ε, πώς θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συνενετική ε, θέση του Κοινοβουλίου προς την πρόταση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Σε αυτή την περίοδο της κρίσης υπάρχουν συνάδελφοι που θεωρούν ότι για να ε, προσδιορίσουμε ένα πολιετές ε, πρόγραμμα υγείας βρίσκουμε ένα πρόσφορο τρόπο να καλύψουμε τις ανησυχίες ε, μεγάλου αριθμού πολιτών ε, και να δώσουμε μια απάντηση ως προς το ρόλο που θα διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζω, Πρόεδρε, και πάλι ότι πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Αυτό το πρόγραμμα οπωσδήποτε θα πρέπει να συνιστά προσθέμενη αξία σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα στον τομέα της υγείας. Συμφωνώ και σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή όλους. Συμφωνώ λοιπόν για αυτό για το οποίο και εσείς επιμείνατε, δηλαδή ε, για το θέμα της ισότητας ε, των πολιτών ενώπιον ε, του συστήματος υγείας. Αυτό το επαναλαμβάνουμε, είναι η μόνιμη εποδός μας τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα σε αυτή την περίοδο της κρίσης αποκτά νέα σημασία, διότι με την κρίση που υπάρχει σε διάφορες ε, χώρες έχουν γίνει σοβαρές περικοπές στον προϋπολογισμό της υγείας άρα θα πρέπει να αγωνιστούμε για να ε, διατηρήσουμε τα κονδύλια. Ε, επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε να συνοδεύσουμε τον Επίτροπο Νταλή σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να διατηρηθούν τα κονδύλια και ήδη έχει πετύχει μια αύξηση του προϋπολογισμού. Ας μην χαθεί λοιπόν αυτή η αύξηση μέσα στον έφος των συζητήσεων. Επιμένετε πολύ στην πρόληψη. Αληθεύει αυτό. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την υγεία των ε, πολιτών και θέλουμε να ε, προσφέρουμε μία προσθέμενη αξία για τους πολίτες και για την Ένωση, ε, ε, συνειδητοποιούμε ότι οι υγιείς πολίτες σε κάθε περίπτωση είναι ό,τι θετικότερο έχουμε να κάνουμε για την οικονομία μας. Λοιπόν, αυτά τα σημείωσα, σημείωσα και όλες τις επιμέρους παρατηρήσεις σας για να καταλάβω με ποιο τρόπο θα μπορέσω να ενσωματώσω αυτές τις παρατηρήσεις καθώς και τις μελλοντικέ αστροπολογίες στο σχέδιό μου. Θα συνεχίσω δε στενή συνεργασία με όλους σας, ευελπιστώντας να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική Συμφωνία. Για τον τίτλο, ε, ναι, εντάξει, συνειδητοποιώ ότι όλοι επιθυμούν τροποποίηση του τίτλου. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, ούτω ώστε ε, και μέσα από τον τίτλο να διαβιβάζεται ένα ε, εύληπτο ε, μήνυμα ε, προς τους πολίτες, ώστε Ε, ε, οι εξελίξεις να μην είναι επιζήμιες ε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που δεν κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο, τους εκπροσώπους τους δηλαδή, που παρενέβησαν και σχολίασαν την έκθεσή μου. Είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων για τη μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κροσέτ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Είπαμε ότι είναι η 16η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, ενώ τον Ιούνιο στις 20, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας Επιτροπής, θα ψηφίσουμε εδώ την έκθεση και έχει σχέση ε, μετά και το πώς θα προχωρήσουμε στην Ολομέλεια. Αυτό δηλαδή έχει σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές, όπως και πολλά άλλα άλλωστε επηρεάζονται από αυτό καλή συζήτηση και ένα από τα σημεία ε, επίκρισης είναι η επικεφαλίδα ε, του προγράμματος και ανάλογα με τη γλώσσα μπορεί να ε, οδηγεί σε παρεξηγήσει παρεμηνίες, αλλά και το περιεχόμενο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το πρώην έξι, αν θυμάστε, του κυρίου Πυρίλο. ειδικέ διατάξει σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το στόχο επενδύσει στην ανάπτυξη και την απασχόληση και για την κατάργηση του κανονισμού 1080 του 2006. Ο κύριος Πυρίλο, παρακαλώ. Εισαγωγικά. Έχουμε ένα τέταρτο για την έκθεση αυτή. Να είστε σύντομοι, παρακαλώ, γιατί έχουμε και εκθέσει κυρία Σοκονή. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και πολύ σαφής. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μεταθέσατε τη σήμερα γιατί χτες, ε, όπως ξέρετε, είχα διάφορες υποχρεώσεις λόγω των εκλογών που είχαμε στην Ιταλία. Κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο πρότασης της ε, Επιτροπής ε, που παρουσιάζει τη νέα περιφερειακή πολιτική το περιβάλλον ε, και η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά τα δύο είναι ένα σημαντικό τμήμα της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η πολιτική συνοχή είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για να στηριχθούν διάφορα τμήματα των προγραμμάτων και των επενδύσεων έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια οικονομία με περιορισμένες ε, εκπομπές διοξούδιου διοξιδίου άνθρακα. Η πρόταση αυτή για την περιφερειακή ανάπτυξη ε, προβλέπει βέβαια ε, μία προσαρμογή της ε, τάξης του 6%. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν επαρκεί λόγω του ότι ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος. Για το λόγο αυτό εγώ έχω καταθέσει μία πρωτοβουλία που αυτό το 6% θέλω να το αυξήσουμε στο 10%. Επίσης, ανάμεσα στους ε, θεματικούς στόχους αναφέρω και τις ε, προτεραιότητες που περιλαμβάνει το άρθρο 5, παράγραφος 6, εκεί όπου γίνεται λόγος για την προστασία του περιβάλλοντος και για την επάρκεια των πόρων. Οι περισσότερες τροπολογίες αφορούν το παράρτημα υπαριθμών 1, δηλαδή ε, κοινού δείκτες για τον, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κυρίως για την πρόληψη κινδύνων που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουμε μια ε, οικολογική συστημική προσέγγιση. Είναι σωστό να υπάρχουν κοινοί δείκτες για την βιοπικιλότητα και να, λαμβάνονται, να λαμβάνεται υπόψη ε, και ο θαλάσσιος πλούτος. Επίσης, να λαμβάνεται υπόψη ε, και η προστασία των παράκτειων και θαλάσσιων ενδιαιτημάτων. Νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να βελτιώσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση γιατί τα κρατημέλη, τους μόνους πόρους που έχουν είναι οι κοινοτικοί πόροι με ιδιαίτερη αναφορά ε, στις ε, περιφέρειες που έχουν σχέση με τον στόχο που σας ανέφερα. Και θα είμαι βέβαια στη διαθεσία και ανοιχτός για σχόλια και προτάσεις που μπορούν να γίνουν από τους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, δίνω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Παρακαλώ. Η κυρία Γιούζο. Η κυρία Γιούζο χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Έλεγα ότι θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Το πρώτο που έχω να πω ότι τα κονδύλια αυτά ήταν ένα σπουδαίο μέσο στο παρελθόν και ελπίζω να συνεχίσουν και στο μέλλον να διατηρηθούν για την ανάπτυξη των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τις ε, γραμμές που δεν πρέπει να επιδοτηθούν και με τους στόχους και με τα ποσοστά που προτείνονται σε σχέση με τον κύριο Πυρίλο να του πω ότι έχει κάνει σπουδαία δουλειά. Στροπολογίες μόνο να πω. Κάπου προτείνει να συμπεριληφθεί ε, το σημείο 6 του άρθρου 9 του κανονισμού, του οριζόντιου, προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ σε αυτό, αλλά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλοι, όχι μόνο ορισμένοι. Επίσης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιφέρειες ε, προτείνει να συμπεριφθεί το σημείο 6 και συμφωνώ, αλλά αν είναι σε τόσο μειονεκτική ε, θέση. Δεν χρειάζεται να συμπεριφθεί το σημείο 6, να το αφήσουμε στο σημείο α. Το ποσοστό τώρα, να περάσουμε από το 6% στο 10%. Για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αυτό είναι πολύ υψηλό ποσοστό, γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Νομίζω θα πρέπει να αφήσουμε περισσότερη ευελιξία και περιθώριο στις περιφέρειες της ίδιας να αποφασίσουν ποιες είναι οι ανάγκες. Δεν συμφωνώ να αυξηθεί αυτό στο 10% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, θα το άφηνα στο 6. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ ισορροπημένη. Για τους δείκτες, τους κοινού που θέλει ο εισηγητής, βεβαίως και θα πρέπει να ορίζονται με τρόπο σαφή, δεν ε, αμφιλέγω, αλλά χρειάζεται υποδομή αυτό και έχει κόστος. Έτσι, δεν θα πρέπει να είμαστε πάντα εξαντλητικοί σε αυτούς τους δείκτες, ούτε να θεσπίσουμε νέους, γι' αυτό σημαίνει κατασπατάληση πόρου και δεν έχουμε ούτε πόρους ούτε χρόνο γι' αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Γιούσο. Από τους φιλελευθέρους η κυρία Μάνε. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ καλό το σχέδιο γνωματότησης. Τα περισσότερα μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και για τις τροπολογίες. Ήταν καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα θέματα του περιβάλλοντος στο ΜΕΝ και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχω μερικές λεπτομέρειες ε, ως παρατηρήσεις για τις τροπολογίες. Είναι πολύ καλό αυτό το θέμα ε, της ανακύκλωσης των αποβλήτων. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, συγκοινωνίες. Ε, το άλλαξε, ε, δεν μιλάει για αστικές ε, συγκοινωνίες, αλλά για δημόσιες συγκοινωνίες και μπορώ να το υποστηρίξω. Για το ποσοστό αυτό που αυξάνεται από 6 10% και εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Καλό είναι οι λιγότερο επιτυγμένες περιφέρειες να επενδύουν σε θέματα περιβαλλοντικά και να λαμβάνεται αυτό υπόψη από το Τομείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά το 6% νομίζω αρκεί. Επίσης, οι δείκτες θα πρέπει να ορίζονται σαφώς και να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή ξεκάθαρα, γιατί μέχρι τώρα μας τα λέει λίγο αόριστα τα θέματα αυτά των δικτών. Θεματικές προτεραιότητες είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη προγραμματική περίοδο της ε, περιφερειακής πολιτικής και είμαι βέβαια ότι θα το συζητήσει αυτό και η Περιφερειακή Επιτροπή και καλό είναι να γίνει ευρύτερη συζήτηση στην Περιφερειακή. Ωστόσο δεν θα πρέπει να διευρύνουμε πάρα πολύ το πεδίο γιατί θα είναι αντιπαραγωγικό να θέλουμε να βάλουμε σε αυτή την έκθεση τα πάντα. Πάντως είναι καλή βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγελος, τελευταίος παρόν σκιώδης. Σωστά το είπα τώρα, Χρυσόγελος. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση για το Περιφερειακό Ταμείο είναι σε μια σωστή κατεύθυνση αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε σε πιο φιλόδοξου στόχους ό,τι αφορά τα ποστά χρηματοδότηση που αφορούν ε, την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιοπικιλότητα. Ε, πρέπει να ε, πετύχουμε την εφαρμογή τη στρατηγικη Ευρώπη 2020 και των στόχων που θέτει και γι' αυτό νομίζουμε ότι το κεφάλαιο 3 δεν πρέπει να απαγορεύει καινοτόμε επενδύσει σε αναβάθμιση των υπηρεσιών των οικοστημάτων, σε πράσινε υποδομέ. Στι φιλικέ προ το περιβάλλον μεταφορέ, στην προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση τη βιοπικιλότητα, στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων όσον αφορά και στι πιο πλούσιε και αναπτυγμένε περιφέρειε. Δηλαδή θέλουμε μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερική ανάπτυξη, στου τομεί του περιβάλλοντο και των μεταφορών να ενισχυθούν οι πράσινε καινοτομίε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια στρατηγική συνεκτική Α μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ακόμα και στι ε, πλούσιε και αναπτυγμένε περιφέρειε υπάρχει τεράστιο έλλειμμα και επενδύσεων αλλά και παρέμβαση σε αυτού του τομεί. Και ιδιαίτερα ακόμα και μέσα σε αναπτυγμένε περιφέρειε υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα, υπάρχουν περιοχέ που δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένε στο σύνολο μια περιφέρεια και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και εκεί, σε αυτέ τι περιοχέ που στο εσωτερικό μια αναπτυγμένη περιφέρεια παρουσιάζουν υστέρηση. Και νομίζω ότι κυρίω οι καινοτόμε περιβαλλοντικέ παρεμβάσεις είναι αυτέ που λείπουν. Σε ό,τι αφορά του στόχου για τι κλιματικέ αλλαγέ, θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πιο φιλόδοξε δεσμεύσει για εξοικονόμηση ενέργεια και ανανεώσιμε πηγέ μέχρι το 2020 και γι' αυτό προτείνουμε να αυξηθεί το ποστό χρηματοδότηση για του κλιματικού στόχου για τις πιο αναπτυγμένες και τις μεταβατικές περιφέρειες από το 20% σήμερα που προτείνεται στο 25% ενώ αντιστοίχως και για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές να ανέβει ο στόχος από το 6% στο 15%. Στα άρθρα 4 και 5 ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να δυναμώσουμε την πρόταση της Επιτροπής και την έκθεση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε επίπεδο οικοστημάτων και βιοπικιλότητας για να δυναμώσουμε το φυσικό κεφάλαιο και τις παραγωγικές υπηρεσίες των οικοστημάτων αλλά και για να προσαρμοστούμε πιο αποτελεσματικά στι κλιματικέ αλλαγέ και να τι αντιμετωπίσουμε προληπτικά, δημιουργώντα παράλληλα και νέε θέσει εργασία. Τέλο, τα παραρτήματα πρέπει να βελτιώσουμε του προτινόμενου κοινού δείκτε. Είναι σημαντικό αυτοί να ανταποκρίνονται ε, στου στόχου Ευρώπη 2020 και στι ε, έννοιε για βιώσιμη ευημερία. Δηλαδή, ε, δεν μπορούμε να μετράμε μόνο χιλιόμετρα, δεν μπορούμε να μετράμε μόνο ε, αριθμό κατοίκων, αλλά να έχουμε σωστούς δείκτες ακόμα και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, και της πρόληψης των κινδύνων, θα πρέπει να έχουμε μαζί με την πολιτική προστασία και δείκτες που μετράνε την αύξηση ικανότητας πρόληψης και αντοχής των οικοστημάτων και μείωση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται απολύτως με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Vielen Dank. Der Vertreter der Kommission... Ευχαριστώ. υποχρεώθηκε να πάει στην Περιφερειακή Επιτροπή για ε, μια συζήτηση άλλη, γιατί αλλάξαμε τη σειρά των θεμάτων. Είναι δικαιολογημένα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να δώσω το λόγο στον εισηγητή, αλλά προηγουμένω σε άλλου δύο. Πρώτα στον Πέτερ Λίζε και μετά στη Σοφία Κονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βέβαια θα είμαστε σύντομοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι η Επιτροπή περιβάλλοντο εμεί θα πρέπει να υποστηρίξουμε πολύ τον Επίτροπο κύριο Χάν. Για πρώτη φορά τίθεται αυτό το θέμα του περιβάλλοντο προστασία ε, του κλίματο και ενεργειακή απόδοση στα περιφερειακά και εμεί θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Και για λόγου πολιτικού έχει νόημα να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως προτείνει ο εισηγητής να αυξήσουμε και τα ποσοστά γιατί προτάσεις για περικοπές έρχονται ε, αρκετές από τα κράτη-μέλη και ίσως και από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Μια που κάνει αυτή την προσπάθεια ο Επίτροπος, καλό είναι εμείς να τον υποστηρίξουμε και έχει δίκιο ο εισηγητής. Μια δική μου πρόταση, αν επιτρέπετε, στον κανονισμό μέχρι σήμερα, ο υφόρος τουρισμός είναι προτεραιότητα. Δυστυχώς χάθηκε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι παρόλα αυτά μπορούν να συνεχιστούν τα προγράμματα και ο υφόρο τουρισμό είναι όμως ε, και η δική μας προτεραιότητα στην Επιτροπή μας και θα αισθανόμουν πιο ε, ήσυχο ε, αν διατηρηθεί, γιατί επί τόπου μπορεί κανείς να το παρεξηγήσει και θεωρεί ο κόσμος ότι θα σταματήσουν τα προγράμματα, ενώ δεν πρέπει. Ευχαριστώ, κυρία Οκονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της εργασίας που επιτέλεσε. Όπως είπε και ο Πίτερ Λίζε, πρέπει να υποστηρίξουμε τον Επίτροπο Χάνας στις προσπάθειες που θέλει να κάνει για αυτό το τόσο σημαντικό για το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα θέμα. Σε σχέση τώρα με ε, την εστιασμένη θεματοποίηση για τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Ε, μιλήσαμε για τροποίηση του ποσοστού, αύξηση στο 6% και δεν θέλω να περιοριστώ σε αυτό. Στο άρθρο 3 θα πρέπει να διαγράψουμε την παράγραφο όπου αναφέρεται ότι οι επενδύσεις που βελτιώνουν τις βασικές υπηρεσίες προς τους πολίτες απαγορεύονται. Γιατί, Γιατί να απαγορεύσουμε τις βασικές υπηρεσίες προσφέρονται στους πολίτες, τώρα τις χρειάζονται ακόμη περισσότερο λόγω της κρίσης. Χρειάζονται υποστήριξη, βοήθεια, συνδρομή. Πρέπει να διαγράψουμε αυτή, την αράδα. Όπως ε, ήδη έχει τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω διαφόρων ψηφισμάτων, κάποιες υποδομές, όπως παραδείγματος χάρη υποδομές για την υδροδότηση, δεν έχουν τελειοποιηθεί ως προς την εδαφική κατανομή ε, και των δικτύων ε, στην εθνική επικράτεια, σε κάποια κράτη-μέλη ε, και κάποια κράτη-μέλη μάλιστα δεν είναι πλέον επιλέξιμα για τις επιδοτήσεις του ΕΤΠΑ με στόχο την μόχλευση ως προς την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών αυτών. Οπότε σε χωροταξικό επίπεδο θα πρέπει να επιδιωχθούν ποιοτικά και σε υποδομές, κυρίως στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και κράτη-μέλη. Να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη λοιπόν στο σχεδιασμό και θα συνεχίσουν μόνο στη συνέχεια. Ας περάσω τώρα στην έρευνα και την καινοτομία. Ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μια πραγματική προσπάθεια αποτελεσματική. Ε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται με, τους, ε, με τον εξοπλισμό για ε, να γεμίζουν ευκολότερα και σε διάφορα σημεία πρόσβαση σε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για τον αθλητισμό τώρα, συνιστά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ο αθλητισμός είναι ένα μέσο αναβάθμισης της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει να καταστήσουμε δυνατές λοιπόν τις επενδύσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ε, το οποίο συνιστά πρόβλημα σε όλα τα κράτη, σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις και δεν ενθαρρύνουμε έτσι τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτό το τόσο πολύτιμο ε, μέσο δημόσιας υγείας. Ο κύριος Πυρίλο έχει το λόγο, εισηγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, πολύ λίγα πράγματα θα πω. Καταρχήν θέλω να ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που κατόρθωσα να προκαλέσω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ε, δεν ε, είπα ότι θα τα εξετάσω όλα. Ε, αντίον... Ε, είπα ότι είμαι ανοιχτό ε, στις ε, παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων. Όσον αφορά λοιπόν στις ε, τροπολογίες που θα συζητήσουμε, θα τις συζητήσουμε αυτές για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πλέον την αρκετά ενδιαφέρουσα δυνατότητα που μας προσφέρεται από την Επιτροπή να επανεξετάσουμε έναν κανονισμό. Γι' αυτό λοιπόν ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια αυτή η δυνατότητα και αυτή η ρύθμιση να εφαρμοστεί και στα 27 κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι Μαΐου στις 12 ε, η ώρα. Θα ψηφίσουμε στις 21 Ιουνίου για την τροπολογία και στην ε, Επιτροπή Περιφερειών η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούλιο και μετά από ό,τι φαίνεται το όλο θέμα θα πάει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου μετά τις θερινές διακοπές. ευχαριστούμε πάρα πολύ πολύ για όλα αυτά που είπατε και πάμε τώρα και πάλι στην ημερήσια διάταξη στο σημείο υπαριθμών 18. Ε, εκεί είναι η έκθεση της κυρίας ε, Σοφή Οκονή στην οποία θα ήθελα και να δώσω το λόγο. Παρακαλώ κυρία Οκονή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι έχουμε ήδη κάνει την ανταλλαγή απόψεων και την πρώτη συζήτηση για αυτή την έκθεση. Αυτό το νομοθετικό πακέτο καλύπτει τρεις βασικούς στόχους. Ενθάρρυνση ε, της πρόοδου στο σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης βοηδών για τους ε, εκτροφείς που θέλουν με προαιρετικό τρόπο να το ε, εφαρμόσουν. Δεύτερον, ε, παράλληλη ανάπτυξη τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφυγή μάλλον της παράλληλης ανάπτυξης ε, τεχνολογιών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτον, αποφυγή επικαλύψεων και ε, ομοιόμορου Κανόνε για όλου του εκτροφείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει κλείσει το φάκελο, αλλά θα ήθελα να σα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή για αυτό το νομοθετικό πακέτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τι δύο προτάσει τη ε, στι 30 ε, Αυγούστου πέρυσι, δύο νομοθετικέ προτάσει. Διορίστηκα εισηγήτρια τον Οκτώβρη του 2011 και κατέθεσα τις προτάσεις μου τελικά τον Ιανουάριο του 2012. Ε, μετά από μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Επιτροπή Γεωργίας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, σχεδόν για έξι μήνες ε, διεκόπη η διαδικασία. Στις 4 Απριλίου του 2012 δημοσίευσε τροποποιητική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τελικά έχει την αρμοδιότητα η Επιτροπή Περιβάλλοντος. ε, ε ξαναλέω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε αναθεωρημένη πρόταση ε, και γι' αυτό το λόγο προτείνω να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει τις αλλαγές που επέφερε στην πρότασή της για να συνεχίσουμε μια, με μια κοινή συζήτηση επί της αναθεωρημένης πρότασης. Πιστεύω ότι... Ε, ε, θα μπορούσαμε να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει τα νέα στοιχεία πρώτα και μετά συνεχίζει η συζήτηση. Πρόεδρος μας, σας ακούσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Οκονή, την εισηγήτρια, που μας δίνει την ευκαιρία να εξηγήσουμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές ε, αληθεύουν όλα αυτά που σας είπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως είχε καταθέσει την αρχική πρόταση που ενέκρινε το Σώμα των Επιτρόπων τον Αύγουστο του 2011 και στη συνέχεια λάβατε όλοι μια νέα ε, αναθεωρημένη πρόταση τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Θα ήθελα να σας ε, παραθέσω τους λόγους ε, που αιτιολογούν αυτήν την αναθεωρημένη πρόταση, μειώνοντας, ελπίζω έτσι, τις ανησυχίες που εκφράζουν τα μέλη της Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, η αρχική πρόταση, η οποία εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2011, είχε μεταξύ άλλων το στόχο να εξασφαλίσει ισότιμους όρους για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί ε, αναγνώρισης και επισήμανσης ε, των ε, βοηδών. Βάσει του άρθρου 22 της αρχικής πρότασης προβλέπονταν ίσοι όροι μέσω μόνο πράξεων, εκτελεστικών πράξεων. Στη συνέχεια όπως προβλέπετε στο άρθρο 22, οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκριναν ενδεδειγμένο να ε, καταθέσουν νέα πρόταση ε, προσπαθώντας να εξηγήσουν τις νέες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και εισαγάγοντας ε, μια νέα αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης των πράξεων εξουσιοδότηση συμπληρώνοντας έτσι την αρχική διάταξη περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Εξήγησα λοιπόν αρχίζοντας τώρα τη την ε, νομική προσέγγιση του ζητήματος και η τελευταία πρόταση, η αναθεωρημένη πρόταση που θα είναι και η βάση των μελλοντικών ε, διαθεσμικών διαπραγματεύσεων προβλέπει στο άρθρο 22 παράγραφος 3 τροποποίηση με βασικό στόχο να συμπληρώσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέποντας και πράξεις κατεξουσιοδότηση πέρα από τις εκτελεστικές πράξεις. Ξέρετε ότι στο διατακτικό κάθε ε, νομοθετικής πράξης πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή με τις αιτιολογικές σκέψεις. Άρα τροποποιήσαμε και δύο εκτιμώντα, δύο αιτιολογικές σκέψεις. Το μόνο λοιπόν που κρύβεται πίσω από την αναθεωρημένη πρόταση Επιτροπής είναι αύξηση της αρμοδιότητας ε, της Επιτροπής για το άρθρο 22, για τις κυρώσεις δηλαδή. Τίποτε άλλο δεν κρύβεται πίσω από τη νέα πρόταση και θα ακούσουμε πολύ ευχαρίστω τα σχόλια και τις προτάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους και οδησίγητες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. Κυρία Οκονή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφος επανέλαβε αυτό το θέμα της αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της ε, δυνάμωσης, το empowerment. Θα σας έδινα και μια πολιτική υπόδειξη στις κατοξιοδότηση πράξης, παρακαλώ να αναφέρεστε και στο Κοινοβούλιο και στο ρόλο του. Θα σας ε, συμπαθούν και περισσότερο ορισμένοι. Η τεχνική ε, αλλαγή που προτείνεται με ΑΙ είναι κάτι το οποίο εγώ θα συζητήσω στην ομάδα μου να το εγκρίνει. Ε, αναλύω ότι το είπε και η κυρία Κονή. Τα βασικά σημεία θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε το θέμα της ηλεκτρονικής σήμανσης, της υποχρεωτικής μάλιστα, μια μεταβατική ρύθμιση ενδεχομένως να βρεθεί και το θέμα της συνέχισης της δυνατότητας ε, εθελοντικής σήμανσης στα κράτη-μέλη. Κάτι που μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει και το περιεχόμενο του κανονισμού. Το απόγευμα θα ψηφίσει η Επιτροπή Γεωργίας, ε, τη Σοφία της ελπίζω, ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια σωστή δουλειά. Η μόνη αλλαγή που μας απασχολεί σήμερα με βρίσκει σύμφωνη, δεν έχω να πω τίποτα για το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σύμβασης και της εθελοντικής. Έχω να πω πολλά. Ευχαριστώ. Η Ρίκα Μάνα, επόμενη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη δική μας άποψη, η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή και συμφωνώ όσον αφορά την ηλεκτρονική σήμανση. Πιστεύω ότι ε, πρέπει να είναι σαφές ε, ποιοι είναι οι στόχοι που επιδιώκουμε. Κατόπιν τούτου, ε, εγώ στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά την προαιρετική σήμανση, Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν, όπως σας είπα, είναι καλή. Διότι όλοι αυτοί οι ορισμοί βασίζονται στην ε, κείμενη νομοθεσία, σε αυτά που ισχύουν τώρα. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω να υπάρχει κίνδυνος και σε γενικές γραμμές συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι βλέπω, λέει ο πρόεδρος, ε, δεν ε, ζητεί κανείς άλλος ε, το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Είκοσι λεπτάκια μου δίνετε, πρόεδρε. Καλά τα λέω. Donc, pour ce qui concerne euh, la nouvelle proposition de... λοιπόν, σε σχέση με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, συμπαρατάσσομαι απολύτως με την Dagmar. Κανένα πρόβλημα. Εγώ πλάγιν που αυτή ακριβώς, εκείνη μάλλον ακριβώς την χρονική στιγμή, 7 μήνες μετά την αρχική πρόταση, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει αναθεωρημένη πρόταση. Ε, Βεβαίω συνειδητοποιώ όπως και οι συνάδελφοι ότι οι πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση ε, ε, υπάγονται σε διαδικασίες που είναι ε, πολύ ευνοϊκότερες για το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν έχω καμία, κανένα λόγο να προβάλλω ενστάσεις. Θα συμφωνήσω λοιπόν με την συνάδελφο για το, την υπόλοιπη έκθεση. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε ε, διότι σήμερα χρησιμοποιήσουμε τις συνεδρίες για να λύσουμε αυτό το διαδικαστικό ζήτημα, όπως είπε η Ντάγμαν. Δεν θα ξανανοίξουμε προθεσμία τώρα για την κατάσταση τροπολογιών. Το έχουν συμφωνήσει οι σκιοδησίγητες. Θα δούμε ε, πότε θα ψηφίσουμε τότε στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για τη συγκεντρωμένη και μεθοδική δουλειά. Ήταν πολύ μεγάλη συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλό σημερινό διάλειμμα και το αργότερο αύριο στην Ολομέλεια θα τα ξαναπούμε. Καλή σας όρεξη.